Dear ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κοινή μας συνεδρίαση. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κηρύσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Ρέτζι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Κότερ της Επιτροπής των Περιφερειών. Αγαπητέ κύριε Κατάινεν, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ρέτζι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Υποεπιτροπή Κοτέρ αυτής, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να σας καλωσορίσω όλους θερμά επί τη ευκαιρία αυτής της κοινή ακρόασης για την εφαρμογή της αστικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σκοπός της συνεδρίασης είναι να ενθαρρύνει ε, την Ευρωπαϊκή Αστική Ατζέντα, την ατζέντα για το άστι, για τον αστικό χώρο. Ο κύριος Πέρκλε και η κυρία Βέστφαλ έχουν συντάξει έγγραφα με βάση κοινέ ιδέες και κοινέ προτάσεις. Και πιστεύω ακραδάντως ότι όλα τα μέλη και της ΡΕΤΖΙ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΚΟΤΕΡ της Επιτροπής των Περιφερειών απαιτούν συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον αστικό χώρο. Πέρσι το Σεπτέμβριο το Κοινοβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμά του για τις αστικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Χωροτακτικής Πολιτικής με μεγαλύτερη εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση μια νέα μέθοδο διακυβέρνησης πολλαπλών επιπέδων. Θα έχουμε μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης έτσι ώστε οι ΟΤΑ να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τις αρχές της αναλογικότητας και επικουρικότητας ενώ στο ψήφισμα υπογραμμίζεται επίσης ότι πρέπει να έχουμε την καλύτερη δυνατή μόχλευση από τα επενδυτικά κεφάλαια με συνέργειες μεταξύ ευρωπαϊκών ε, και εθνικών προγραμμάτων και χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε ακούσει τις παρουσιάσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, η οποία στηρίζει αυτή τη διαδικασία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και κατά τη διάρκεια της, ε, Ιρλανδική, της Ολλανδικής Προεδρίας θέλει να υπάρξει το σύμφωνο του Άμστερνταμ για βελτίωση του νομοπαρασκευαστικού έργου, για αξιοποίηση και βελτίωση των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων και για δημιουργία μιας πλατφόρμας γνώσης για τον αστικό χώρο. Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες της Ολλανδικής Προεδρίας και θα εκφέρουμε τη θέση μας ως Κοινοβούλιο στο, σε σχέση με το τελικό κείμενο του Συμφώνου του Άμστερνταμ, το οποίο περιμένουμε το Μάιο από την Ολλανδική Προεδρία. Ε, το σημαντικό βέβαια είναι να έχουμε νέες μεθόδους εργασίας να έχουμε εταιρικέ σχέσει και κοινή αξιολόγηση αντικτύπου τη νομοθεσία Για να πετύχουμε αυτού του στόχου χρειαζόμαστε μια πρακτική και συγκεκριμένη προσέγγιση, η οποία θα αντικατοπτρίζει τι ανάγκε που, που υπάρχουν επιτόπου και η οποία θα αντικατοπτρίζει και την εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων επίπεδων διακυβέρνηση, Οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι μέρο του παγκόσμιου συστήματο στον κόσμο και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μα κάθε φορά που προετοιμάζουμε την ατζέντα για το Habitat Free, για το τρίτο ενδιέτημα. Και θα πρέπει η δική μας ατζέντα να είναι πλήρως συμμορφούμενη και συντονισμένη με τους στόχους της παγκόσμιας ατζέντα για τον αστικό χώρο. Και ελπίζω η σημερινή ακρόαση να συμβάλλει στο να εμπλουτίσουμε την κατανόησή μας για όλα αυτά τα θέματα, να ακούσουμε τους ερευνητές, τους εμπλεκόμενους φορείς, ε, τους θεσμούς, τα ιδρύματα που δραστηριοποιούν δραστηριοποιούνται επί τόπου. Στόχος μας είναι η ατζέντα αυτή επιτέλους να αρχίσει να εφαρμόζεται, να τεθεί σε κίνηση και σίγουρα όλοι συμμεριζόμαστε αυτή τη βούληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κατάινεν για να κάνει και εκείνος κάποιες ε, εναρκτηρίες παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Κατά νέο. Με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία λόβα. Κυρία Πρόεδρε της Υποεπιτροπής της Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ρέτζι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάδελφοι από την Επιτροπή Κοτέρ της ε- ε- Επιτροπής των Περιφερειών, μέλη του προσωπικού κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Μιχαηλόβα και τα μέλη της ΡΕΤΖΙ γιατί δέχθηκαν την πρότασή μας να παραστούμε όλοι στη διοργάνωση αυτής ε, της κοινή ακρόασης και αυτό δείχνει πόσο δεσμευμένοι είμαστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια νέα αστική ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο ε, υπόθηκε στην κοινή μας δήλωση ε, με τίτλο «Στην πορεία προς το σύμφωνο του Άμστερνταμ», δήλωση που δημοσιεύσαμε το περασμένο Οκτώβριο. Η πολιτική συμμαχία μεταξύ της Επιτροπής Ρέτζη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Κότερ της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είναι μια εταιρική σχέση πολύ χρήσιμη, καρποφόρο που θα έλεγα, που επιθυμεί να επιταχύνει την εφαρμογή μιας νέας ευρωπαϊκής ατζέντας για το άστι, ε, προκειμένου να ενισχυθούν οι ΟΤΑ, οι πόλεις, ε, και η συμμετοχή αυτών γενικότερα στην ομοπαρασκευαστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, δηλαδή τη συζήτηση για μια ευρωπαϊκή ατζέντα για το άστι. Αυτή τη συζήτηση στην Ευρώπη την ξεκινήσαμε πρώτη φορά το 1997, σχεδόν 20 χρόνια πριν. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη ανακοίνωση για μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για το άστι. Έκτοτε πολλές ε, πρωτοβουλίες έχουν ανακοινωθεί. Έχουμε το Τζέσικα, το Europact, πολύ γνωστές πρωτοβουλίες. 20 χρόνια μετά όμως, μετά από 20 χρόνια συζητήσεων, δηλώσεων, ψήφισματων, παραμένει απούσα η Ευρωπαϊκή η επαϊκή ατζέντα για το άστι. Και επειδή απουσιάζει, δεν υπάρχει συνέπεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ ε, των ε, προγραμμάτων ενίσχυσης από τη μία και επικούρησης και των διαφορών πρωτοβουλειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την άλλη. Και άλλωστε δεν επιτυχάνουν αυτά αποτελέσματα όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές ακριβώς λόγω αυτού του γεγονότος ότι απουσιάζει μια ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άστι και γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Έχοντας, ο στόχο, λοιπόν, τον... Έχοντας υπόψη μας το στόχο της εδαφική συνοχής, κάτι το οποίο υπάρχει στη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, θα πρέπει θεμελιώδες εργαλείο να θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για το ΑΣΤΗ. Είναι ένα εργαλείο για να ενισχύσει την ε, εμπλοκή των ευρωπαϊκών πόλεων στους, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δηλαδή τη διαδραστική σχέση μεταξύ των δύο. Και αυτά είναι τα δύο πρόσωπα της πολιτικής μας θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των περιφερειών και των πόλεων στην ευρωπαϊκή νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ακρόαση για εμάς. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία να ε, ενισχύσουμε τη στενή συνεργασία που έχει ήδη εδρεωθεί μεταξύ των δύο εξαιρετικών μας εισηγητών. Έχουμε τον κύριο Πάστα Κέκ από την Επιτροπή των Περιφερειών και την κυρία Κίστιν Βίσμαν από την Επιτροπή Ρέτζι. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούν να έχουν καλές συνέργειες και ε, θα μπορέσουν να, ε, να πάνε παραπέρα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σχετικό. Σίγουρα, εάν ε, έχουμε κοινή θέση, θα έχουμε πιο ισχυρή πολιτική θέση ούτως ή άλλως. Και έχουμε και την κυρία Λόπερ, την εισηγήτρια για τη νέα γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία προτείνει συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για το άστι. Και η Ολλανδική Προεδρία έχει αναλάβει το θέμα και πρέπει να υπογραμμίσουμε το ρόλο της Ολλανδικής Προεδρίας και να ταχθούμε υπέρ αυτού του θέματος, γιατί η Ολλανδική Προεδρία το θεωρεί ως προτεραιότητά της. Επομένως βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι δρόντες συνεργάζονται και αυτό είναι πολύ καλό. Και με πολύ μεγάλη χαρά θέλω να υπογραμμίσω και το εξής. Η σημερινή ακρόαση είναι η πρώτη κοινή ακρόαση μεταξύ των δύο υποεπιτροπών μας. Είμαι πεπισμένος ότι θα γίνει μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ αμφωτέρων των μελών μας και αυτό θα είναι μια σημαντική τομή στην κοινή δουλειά που έχουμε για την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άστι. Πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να είναι ισχυρή η θέση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών. Εν ώψη του Συμφώνου του Άμστερνταμ που θα ε, υιοθετηθεί τον Μάιο του 2016. Κάτι το οποίο ελπίζουμε Εάν δούμε τα θέματα που είναι προτεραιότητα για την Ολλανδική Προεδρία και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι το πιο ενδιαφέρον για εμάς είναι π.χ. οι θέσεις απασχόλησης και οι δεξιότητες στην τοπική οικονομία, η αστική φτώχεια, η κοινωνική συνοχή, η κινητικότητα, η συμπερίληψη ή η ένταξη μεταναστών και προσφύγων. Στόχος της ατζέντα είναι να είναι ένα λειτουργικό πλαίσιο να δώσει εργαλεία για να ξεκλειδώσει το δυναμικό των πόλεων, να απελευθερωθεί το δυναμικό των πόλεων και έτσι να έχουν κανόνες οι πόλεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εναρμονιστούν με την ευρωπαϊκή πολιτική. Ξέρετε, σε πέντε χρόνια το 80% των Ευρωπαίων πολιτών θα ζει μέσα σε πόλεις και το 85% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ θα παράγεται μέσα σε ευρωπαϊκές πόλεις. Όλα αυτά δεν απαιτούν μόνο νέα νομοθεσία, νέα χρηματοδότηση και νέες δομές και πεδία αρμοδιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται κατά τη γνώμη μου επίσης και μία νέα μέθοδο εργασίας. Μία ισχυρότερη εταιρική σχέση για θέματα που έχουν να κάνουν με το άστι σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε όλα τα θεσμικά επίπεδα. Μιλούμε για αρμοδιότητα multi-level, πολλαπλών ή διαφορετικών επίπεδων. Έχουμε την οικονομική την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, τον κόσμο της οικονομίας, όλοι αυτοί πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή είναι η γνώμη μου και θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Μιχάλοβα για τη στήριξη ε, την ιδέα για τη διοργάνωση αυτή τη κοινή ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τώρα με τι παρουσιάσεις ε, των προσκεκλημένων μας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όπως συνήθως έχουμε πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τις συνεδριάσεις μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ζητήσω από όλους τους προσκεκλημένους να κρατήσουν τα όρια του χρόνου ομιλία του και να μην υπερβούν τα 10 λεπτά ο καθένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε τι παρουσιάσει με τα μέλη τη Επιτροπή Κοτέρ, τη Επιτροπή των Περιφερειών. Κύριε Κατανέο, έχετε το λόγο να μα παρουσιάσετε τον προσκεκλημένο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαρά μου θα σα παρουσιάσω την κυρία Κριστίν Χάμζα. Όπω γνωρίζετε, η Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε μία μελέτη από την Metis Consulting για το δυναμικό ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένη, ενός ολοκληρωμένου αστικού θεματολογίου. Ζητήσαμε ποσοτικά παραδείγματα, ευρήματα βασισμένα σε γεγονότα έτσι ώστε να ε, μας βοηθήσει στις ε, πολιτικές μας συστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να καλωσορίσω την Κριστίν Χάμσα, της, ε, με τις consulting για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την μελέτη μας. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας πω πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης μας μέσα σε 10 λεπτά. Το σκεπτικό είναι ε, να επικεντρωθούμε σε ορισμένα συγκεκριμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο αστικό θεματολόγιο. Αυτό που κάναμε είναι αυτό που θα σας παρουσιάσω. Βλέπετε το πόσο ε, πολύπλοκο ζήτημα είναι η αστική ανάπτυξη και τον διοικητικό φόρτο που πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, οι διοικήσεις. Υπάρχει αυστηρότητα στην πολιτική, στην τομεακή πολιτική και στην δομή τη διοικητική. Εμείς επικεντρωθήκαμε σε τρεις εγκάρσιες προκλήσεις, την κλιματική αλλαγή, τη δημογραφική αλλαγή και τη μετανάστευση. Και προσπαθούμε, ειδικά το τελευταίο, να το αντιμετωπίσουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε πέντε περιπτώσεις, πέντε κατηγορίες περιπτώσεων, όπου οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Θα δούμε λοιπόν τις περιπτώσεις αυτές και τις δυνατότητες που έχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Έχουμε λοιπόν τρία βασικά, ε, τρεις βασικές κατηγορίες, αστική οικονομία, κοινωνικός ιστός και αποδοτικότητα των πόρων, μετά αστική διακυβέρνηση και τις μεταφορές, κάτι που για μας περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ως προς τα συμπεράσματα, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι όλοι γνωρίζουμε πως οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι πρωτοπόροι στην ανάπτυξη, οδηγούν την ανάπτυξη έτσι λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι το αστικό θεματολόγιο μπορεί να συνεισφέρει στην όθηση ε, της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι από τη μία πρέπει να ασχοληθούμε με τις τομεακές πολιτικές και το πώς οι τοπικές αρχές θα μπορέσουν να ασχοληθούν και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία ε, τις ε, προκλήσεις που έχουν μέσα στα πλαίσια ενός ε, αστικού θεματολογίου. Υπάρχουν κάποια μέσα που ήδη υπάρχουν, γνωρίζουμε όλοι για το ITI για παράδειγμα, για την FEE εξειδίκευση που πιστεύω πως είναι πολύ καλά προγράμματα, έχουν καλή προσέγγιση η οποία μετά μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη. Επίσης το CLLD την ε, τοπική ανάπτυξη βασισμένη στην ε, κοινότητα και να μην ξεχνάμε ότι το αστικό θεματολόγιο είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Δεν είναι καινούργια ιδέα, όμως δυστυχώς ε, παρατηρείται μία στασιμότητα στην εξέλιξη. Αυτό που χρειάζεται είναι να συμπεριληφθούν όλοι οι φορείς από τη βάση προς την κορυφή διότι η έβρεση λύση είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Καταρχάς χρειαζόμαστε μια προσέγγιση βασισμένη στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Δεν μοιάζουν όλες οι αστικές περιοχές μεταξύ τους και δεν μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιήσεις μια λύση για τα πάντα. Έπειτα είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να συμπεριλάβουμε τους, ε, τις βασικές παραμέτρους και την ε, μόχλευση. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε ποιες πολιτικές μπορούν να χαρακτηριστούν, να χαρακτηριστούν ε, software και ποιες hardware. Για παράδειγμα, η έρευνα θεωρείται λογισμικό ε, εντό εισαγωγικών, ενώ οι ε, υποδομές μεταφορών hardware. Αυτές πρέπει να συνδυαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής. Επίσης χρειάζεται συντονισμός από την κορυφή προς τα κάτω σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο και από την άλλη το αστικό θεματολόγιο πρέπει να περιέχει μέσα και εργαλεία έτσι ώστε οι τοπικές αρχές να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ε, στο έπακρο τα μέσα που διαθέτουν προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες ε, της κάθε πόλης. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η δημιουργία ικανοτήτων και να συμπεριληφθεί το γεγονός ότι χρειάζεται περιθώριο ελιγμών. Από την άλλη όμως χρειάζεται και ε, πάταξη της κατάχρησης εξουσίας από τις τοπικές αρχές. Δύο συστάσεις έχουμε κάνει, δύο ομάδες συστάσεων. Η πρώτη, όπως είπα, αφορά αυτήν την εγκάρσια πολιτική που χρειάζεται έτσι ώστε να συντονιστούν οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονα τομεακός προσανατολισμός στις διάφορες γενικές διευθύνσεις και χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και άλλες στρατηγικές στον χώρο της ανάπτυξης. Η πολιτική συνοχής είναι μια πολιτική που πλησιάζει σε αυτόν τον στόχο, χρειάζεται όμως ε, περαιτέρω πρόθεση. Επίσης, οι τοπικές αρχές πρέπει να ενισχυθούν με τον κατάλληλο τρόπο και το αστικό θεματολόγιο πρέπει, όπως είπα και πριν, να είναι μια πλατφόρμα όπου αυτό θα είναι δυνατόν σε διοικητικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο εντός 10 λεπτών να σας εξηγήσω τις λεπτομέρειες αυτού, όμως ε, εν συντομία χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Η Επιτροπή των Περιφερειών, για παράδειγμα, θα μπορούσε να κάνει μια εντελεχή ανάλυση, να δημιουργήσει διάφορες ομάδες εργασίας, έτσι ώστε να εντοπίσει διάφορες βασικές παραμέτρους, ε, πέρα από τις δικές μας, και να κάνει δυνατή την ε, παρακολούθηση διαφόρων ε, περιπτώσεων που θα οδηγήσει στην δημιουργία συστάσεων. Πρέπει να καταλήξουμε σε μία δέσμη μέτρων που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις σε, αυτά, σε αυτές τις κατηγορίες που σας ανέφερα πιο πριν. και τα κράτη-μέλη εν συνεχεία θα μπορέσουν να αντλήσουν από αυτήν την ε, δεξαμενή μέσων και προτάσεων για να χρησιμοποιήσουν τις ε, κατάλληλες προτάσεις στις δικές τους περιπτώσεις. Η μελέτη είναι αρκετά μακροστοκελής, όποιος θέλει όμως ε, μπορεί να την διαβάσει. Σας ευχαριστώ πολύ. 150 σελίδες είναι η μελέτη σας και αναγκαστήκατε να την παρουσιάσετε μόνο σε 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την παρουσίαση. Τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, καθηγητή Μάικλ Πάρκινσον, ο, οποίος είναι αντιπρίτανης στο, ε, στη Σχολή Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και επίσης είναι εκτελεστικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Πολιτικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Επίσης είναι σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Πάρκινσον θα μας μιλήσει για την αστική πολιτική και την ε, αναζωογόνηση. Έχετε το λόγο κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη μου χαρά που εδώ γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Άρα είναι σημαντική μέρα, σημαντικές στιγμές για τις πόλεις στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα με κάνουν να αισθάνομαι πιο γέρος. Γιατί την Λευκή Βήλο του 97 για τη Βιέννη εγώ την συνέγραψα και επίσης την πρωτοβουλία του 94 για τις πόλεις. Επίσης αντίστοιχη μελέτη του 2005 για την Ολλανδική κυβέρνηση. Έχουμε τώρα αυτέ τι διαφάνειες. Ε, σε 10 λεπτά έχουμε αυτές τις 6 ερωτήσεις. Τι να κάνουμε θα περάσει μπροστά σα όλη μου η ζωή σε 10 λεπτά τέλο πάντων για το 6 τι να πούμε τα, ένα, η εμπειρία μου, η άποψή μου ο σκοπό τη πολιτική για τις πόλεις τι πάει να πει μια επιτυχημένη πολιτική και τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε τα τελευταία 20 ετία η Ευρώπη και το πιο σημαντικό θα βοηθήσει το σύμφωνο του Άμστερνταμ πολλές φορές την ιστορία την ε, αγνοούμε, έχουμε κοντή μνήμη, αλλά τα περισσότερα από όλα αυτά είναι γνωστά. Το θέμα είναι κατά πόσον αναλαμβάνει κανείς δράση. Το 1994, επομένως το κείμενο το έγραψα και επομένως ε, αυτή η διαδρομή κρατάει 25 χρόνια. Η άποψή μου σε όλα αυτά είναι ότι ε, ουδέν κενών υπό τον ήλιο. Όλα τα έχουν πει, ξεχάστε την ευρωδιάλεκτο, και εστιαστείτε στην πολιτική, στη διαδικασία, στην εξέλιξη, στην ουσία. Από το 1992 είχαμε ένα βήμα μπρο, δύο βήματα πίσω, ένα σωρό δηλώσεις, διακηρύξεις και πολύ λίγες δράσεις. Χρειάζεται πολιτική βούληση παντού, σε όλα τα επίπεδα. Συνεργασία Κοινοβουλίου, Επιτροπής Περιφυρών. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί αν δεν γίνει αυτό, τι άλλο να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι έχει δείξει πρωτοπόρα στάση, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Το 2015 είδαμε ότι δεν πέτυχε τίποτα και ελπίζουμε κάτι τώρα να πετύχει τώρα. Ε, τέλος πάντων από τη μια μεριά είναι αυτή η πικρή εμπειρία και από την άλλη είναι η ελπίδα. Τι θα πρέπει να γίνει για την πολιτική της πόλης. Η πολιτική αυτή δεν αφορά μόνο την αναγέννηση των πόλεων, δεν αφορά τους φτωχούς, οικοδομισμένες περιοχές, χρειάζεται εν γέννη μια, ένα φρεσκάρισμα και χρειάζεται επίσης και οικονομικές πινελιές οπότε θα πρέπει πρώτα πρώτα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ποιότητα στις πόλεις επίσης θα πρέπει να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε ό,τι κάνουμε και επίσης θα πρέπει να δούμε το σύστημα γενικότερα σε κάποια χώρα συγκεκριμένα στην Ευρώπη και επίσης θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι τα κίνητρα καινοτομία, ανθρώπινο κεφάλαιο Άρα τώρα θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα πράγματα αναπεριοχή. Θα πρέπει να είναι κάτι οριζόντιο και ούτω ώστε όλε μα οι να είναι πιο ανταγωνιστικέ ε, και έτσι να βοηθηθεί η οικονομία μα και κυρίω η ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Οπότε καθώ κανεί διαμορφώνει μια τέτοια πολιτική βλέπουμε ότι το σύνολο του Άμστερνταμ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αλλά πάρα πολλά που χρειάζεται δεν τα φύγει. Λέμε για ε, γειτονιές, ε, τι κάνουμε, τα κοινωνικά, τις ευκαιρίες, ε, ανταγωνισμό, ε, αγορά, τι από όλα αυτά πρέπει να προσέχουμε, τόπους, πρόσωπα, ε, θεσμικές αλλαγές, να καταργήσουμε το παλιό, να φέρουμε το καινούριο, αφορά την περιφέρεια, την περιοχή των πόλεων, αφορά την πόλη καθεαυτή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάτι σαν την πρωτοβουλία ή θα πρέπει να είναι κάτι που έμεσα περνάει και όχι άμεσα γιατί πολλές φορές άλλοι το λένε πολιτεία της πόλης άλλοι αλλιώς τέλος πάντων αυτό που θα πρέπει να κάνουμε να προβληματιστούμε πάνω σε όλα αυτά που σας είπα και συνεχώς αλλάζουμε γνώμη μια το ένα, μια το άλλο κάνουμε και όπως είπε η Πρόεδρος αυτό που χρειάζεται είναι πολύ περισσότερη σταθερότητα στην γραμμή πλεύσης της πολιτικής και απόδοση γιατί μπορεί να έχουμε ένα σωρό σχέδια, προγράμματα αλλά θα πρέπει να δούμε τελικά ποιες είναι οι δυνατότητες σε κάθε επίπεδο. Αλλά όλα αυτά να μην είναι μόνο αέρας κοπανιστός θα πρέπει να σταματήσουμε αυτό το οποίο γινόταν μέχρι τώρα. Τι πάει να πει πετυχημένη πολιτική για τους πολίτες. Σας είπε δυο λόγια συνάδελφος μου. Όλα αυτά σας είναι οικεία. Θέλουμε να έχουμε ολοκλήρωση κάθεται ε, στο Ινωμένο Βασίλειο το λέμε Humpty ε, Dumpty δηλαδή ε, η κυβέρνηση κόβει ένα πρόγραμμα, διαλύει το πρόγραμμα και προσπαθούν να το ανασυνθέσουν οι πόλεις. Άρα είναι περίπλοκα τα πράγματα, χρειάζονται κίνητρα, κίνητρα συνεργασίας, όχι απλώς διακηρύξεις, δηλώσεις προθέσεων, οριζόντια ε, ολοκλήρωση πολιτικής. Να, επομένως, ποια είναι τα συνθετικά αυτής της πολιτικής. Άρα δεν είναι θέμα τόσο πολύ συντονισμού των υπηρεσιών της Επιτροπής, ούτε είναι θέμα μόνο συντονισμού των υπηρεσιών των ε, τοπικών αρχών. Έχουμε τις πρωτοβουλίες, έχουμε τα προγράμματα, όλα αυτά που συνδεθούν με την ευρύτερη γενικότερη οικονομική πολιτική. Να δούμε και την οικονομική πτυχή, την ανταγωνιστικότητα, ε, ανατόπο, ε, να είναι αυτά όλα κοινωνικά δίκαια και να είναι όλα αυτά η φόρα και βιώσιμα. Και όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα. Άρα ε, χρειάζονται και κάποιοι μηχανισμοί υλοποίηση. Έγραψα εκείνη την πρωτοβουλία για τις πόλεις, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στα χέρια μας, αλλά χρειάζονται ανθρώπινοι πόροι, χρηματικοί πόροι κλπ. Και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να εξεύρουμε τους μηχανισμούς που είναι αναγκαία για το μέλλον. Πάντως, αυτό το έχουμε προσπαθήσει πολύ και έχουμε αυτό τον κατάλογο με τις πρωτοβουλίες της χρόνια. Ενωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Δανία, Ιρλανδία, ε, έχουμε το Urban για όλη την Ευρώπη και κοινό παρνωστής είναι ότι όλα αυτά είναι πολύ αξιόλογα, αλλά μηδέν στο πηλίκο. Για σκεφτείτε το καλύτερα. Ε, ε, τον, έχουμε επανεφεύρει τον τροχό και τίποτα. Και όταν είπα ότι χρειάζεται σταθερότητα στη γραμμή πλεύση των πολιτικών μας, δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει συνεχώς να καταργούμε ότι έχει προηγηθεί. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια πετυχημένη πολιτική, θα πρέπει να ορίσουμε ε, ποιοι είναι οι στόχοι και οι προκλήσεις. Και θα πρέπει να δεσμευτούν πολιτικοί και όχι μόνο ε, στα λόγια. Χρειάζεται οικονομική υποστήριξη, χρειάζεται να υπάρχουν φιλοδοξίες, να υπάρχουν προτεραιότητες. Σε κάθε επίπεδο που βλέπουμε μέχρι τοπικό και θα πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση των πρωτοβουλίων με την χρηματοδότηση. Γιατί αυτό είναι το ζουμί. Θα πρέπει να εμπλακεί ο ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι θέμα μόνο βελτίωση ε, ε, τη απόδοση τη κυβέρνηση, τη διοίκηση. Θα πρέπει να εμπλακούν όλοι, χρειάζονται εταιρικέ σχέσει, συνεργασίε ε, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα γι' αυτό, αλλά χρειάζεται και αυτό και διαφάνεια και ε, λογοδοσία και χρειάζεται και αποφασιστικότητα. Όλα αυτά, επομένως, για να αποδώσουν θα πρέπει να εστιαστούμε στην ανταγωνιστικότητα και στην συνοχή και συνέπεια. Και ανατόπο και όσον αφορά τα πρόσωπα. Είπαμε ευθυγράμμιση ε, πόρων και πολιτικών, θέμα κλίμακας και επικράτειας, περιφέρειας χρειάζονται επομένως αυτά. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις συμβατικές σχέσεις ε, πώς θα εμπλακεί ο δημόσιος τομέας διάφορες υπηρεσίες δηλαδή θα πρέπει να μιλούμε για υλοποίηση και δυνατότητες υλοποίησης και επίσης χρειάζεται και μακρόπνοη στράτευση, δέσμευση. Πολύ ωραία. Όλα αυτά χρειάζονται. Μου μένουν άλλα τέσσερα λεπτάκια. Χρειαζόμαστε όμως όραμα, χρειαζόμαστε αποτελεσματικές θεωρικές σχέσεις, στρατηγική προσέγγιση και θα πρέπει να δεσμευτούν και τις υπηρεσίες και να δώσουν τους πόρους. Και επίσης χρειάζεται και ηγεσία και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε εθνικό. Είπαμε, επί μια εικοσαετία έκαναμε δύο θύματα πίσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ρεαλίστρια, αλλά θέλει, ναι, πρέπει να έχει ε, Έγραψα το 2005 αυτό το κείμενο για τις πόλεις και είπαμε ότι δεν είναι το urban τέλειο, αλλά ε, συνδέει τις πόλεις, ε, κρατάει κάποια θέματα στην ε, επικαιρότητα στο επίκεντρο της προσοχής, άρα το urban θέλει περισσότερους πόρους, πρέπει να μεγαλώσει, θα πρέπει να έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα και την συνοχή. Και το πιο σημαντικό που είχα πει τότε είναι ότι αν μπει σε όλες τις πολιτικές του urban θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι περιχαρακωμένοι οι πόροι, ότι εμπλέκονται οι πόλεις, ότι έχουμε επιλέξει τόπους και προτεραιότητες και ότι θα πρέπει οι δημοτικές ε, αστικές αρχές να ελέγχουν, οι δημοτικές αρχές τέλο πάντων, και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν, αλλά δεν γίνανε. Γιατί προχώρησε το Urban, τέλειωσε, αλλά χάθηκε η αιχμή του. Οπότε δεν νομίζω ότι εμπλέκονται όλοι αυτοί που έβλεπε αρκετά, δεν νομίζω ότι έχουμε αρκετέ δυνατότητε, ούτε νομίζω ότι ευθυγραμμίζουν διάφορε επιμέρου υπηρεσίε, ούτε μα στηρίζουν τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή. Άρα, κάναμε μετά προ τα πίσω. Τότε επίση, είπαμε ότι ήταν ένα σκοτσέζικο κοντού τέλο πάντων ε, ήταν απογοήτευση το κείμενο τη Επιτροπή του 2015 γιατί είπαμε αναγνωρίζονται αυτά τα οποία σα απασχολούν, αλλά πάρα πολύ μικρή ανταπόκριση. Μιλούσαμε για το θεματολόγιο τη πόλη, όμω θα πρέπει να μιλούμε για πολιτική, όχι θεματολόγιο. Στο θεματολόγιο ε, είναι κουβέντε. Η πολιτική είναι πράξη. Επομένω, ε, δεν είχαμε αρκετά για τη διακυβέρνηση και για τις δυνατότητες υλοποίησης. Ναι, ναι, πρόεδρε, δύο λεφτάκια ακόμα. Πέραν αυτών, εγώ διατηρώ την αισιοδοξία μου, δεν είμαι απεσιοδοξό. Και θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ ταυτόχρονα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συγκυρία. Σα είπα αυτά στα οποία δεν πήγαμε καλά στο παρελθόν. Για να εστιαστούμε τώρα σε αυτέ τι προκλήσει, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει, εάν το σύμβολο των δεν, δεν είναι εύστοχο, δεν πιάσει τόπο τέλο πάντων, θα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μα αξίζει τίποτα. Νομίζω ότι ε, προκαλεί τα σωστές αντιδράσεις, ε, φέρνει στο προσκήνιο τα πιο σωστά, ζητήματα που πρέπει, ε, προσπαθεί να ενώσει τις διαφορετικές σωματοδοτικές πηγές κλπ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θερμαλόγια, αλλά είναι ότι είναι ευκταίο. Οπότε, αν κάνει όλα αυτά που βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιο από αυτά, τότε θα κάνουμε βήματα πρόοδου. Θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκλήρωση, να βελτιώσουμε τις σημαντικές σχέσεις με τις πόλεις, ε, θα μπορέσουμε να εμπλακούν περισσότερο οι πόλεις ε, και να μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε το πλάνο ε, για το μέλλον, για το 2020 και επίσης λέμε ότι χρειάζεται να εμπλακεί η εθνική κυβέρνηση, να υπάρχει συνεργασία, να εμπλακούν οι πόλεις, εμπλακόμενοι και λίγο όλα αυτά πολύ ωραία όλα αυτά τα λέει γιατί όλα αυτά ε, θα, θα, θα εμπλέξει λέει το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Περιφερειών κλπ. Το θέμα είναι τώρα πώς θα αποδώσει το σύμβολο του Άμστερνταμ. Ρίξτε μια ματιά, τι λέει, επαναλαμβάνει όλα αυτά τα της τελευταίας 20 ετία. Άρα θα πρέπει τώρα να έχουμε περισσότερη πολιτική βούληση από κομισιόν και κράτη-μέλη για να αποδώσει το ε, σύμφωνο και έτσι να δούμε ποιοι είναι οι φραγμοί για την επιτυχία, θα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό και θα πρέπει να αναρωτηθούμε οι συνεργασίες που υπάρχουν, η, αυτή η διευθύνουσα επιτροπή μπορεί να μας οδηγήσει σε μια επιτυχία. Θα πρέπει να βρούμε κίνητρα, να αλλάξει η νοοτροπία, να αλλάξει η συμπεριφορά και επίσης θα πρέπει να εστιαστούμε στο ποιος είναι ο σκοπός μας αλλά και στη διαδρομή για επίτευξη του σκοπού και ποιος τι θα, τι, θα πρέπει να γίνει και όχι τόσο στα τυπικά. Όπως είπε ακριβώ η συνάδελφος, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε τι γίνεται με όλες τις προκλήσεις, όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Πολλά κράτη-μέλη, ξέρετε, έχουν εμπλαϊκή, πόλεις, ε, αρχές και άρα χρειάζεται να είμαστε αρκετά ευέλικτοι αυτό να γίνει πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Όπως σας είπα, πρόκειται για μια καλή αφετηρία. Ε, βέβαια είπαμε από την άλλη μεριά ε, που μας οδηγεί η εμπειρία, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να πιάσει το από αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή κύριο Πάρκισον για την παρουσίασή σας, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πραγματικά προκλητική θα έλεγα. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μάικ Λέρμαν από τη Στοκχόλμη. Στρατηγικός σχεδιαστής για την πόλη της Στοκχόλμης. Θα μας μιλήσει για τις βέλτιστες πρακτικές και την ε, αϊφόρο χρήση γης. Ένα από τα 20 θέματα του θεματολογίου στην εταιρική σχέση που θα αναπτυχθεί στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση γης είναι μια πραγματική πρόκληση. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τις απόψεις του. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ναι, είμαι σχεδιαστής και έρχομαι από μια πόλη και δουλεύω επί τόπου κυρίως, γιατί ασχολούμαι με τη χρήση γης και είναι η βάση για την ανάπτυξη του άστεως η χρήση της γης. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για το τι κάνουμε στη Στοκχόλμη και να μοιραστώ μαζί σας κάποιους προβληματισμούς μας για το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς την ατζέντα για το άστεο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να δουλεύει ο Μάρκερ. Ναι, φαίνεται η διαφάνεια. Εδώ είναι κάποια νούμερα που θέλω να σας δώσω για την ανάπτυξη του άστεως και τις διάφορες χρήσεις γης. Βλέπετε τις προοπτικές για την εξέλιξη του πληθυσμού στις πόλεις από το 1950 μέχρι το 2030. Όλο και θα μεγαλώνουν οι πόλεις και θα αυξάνεται ο πληθυσμός τους. Και έχουμε και την ύπεθρο, από την άλλη, η οποία θα σημειώνει απώλειες, θα συνεχίσει να χάνει ανθρώπους η Ήπεθρος και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν καταρτίζουμε την ατζέντα για το άστι. Η χρήση γης είναι αυτό που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα για στέγαση, για γραφεία, για υποδομές. Το 4% της Ευρώπης σε 26 χώρες καλύπτεται από τεχνητές επιφάνειες, δηλαδή ε, υποδομές, βιομηχανικά, εμπορικά κτίρια, ε, ζώνες οικιστικές, το 4%. Τη Ευρωπαϊκή Υπήρου καλύπτεται από τέτοιου είδου επιφάνειες. Τι συμβαίνει με τις πόλεις. Το είπατε κι εσείς. Πολλές και διαφορετικές οι μορφές των πόλεων, πολλέ και διαφορετικές οι προοπτικές τους. Πολλοί και διαφορετικοί οι τρόποι να αναπτύξουμε μια πόλη. Στο κέντρο βρίσκεται η Ευρώπη. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζουν σε σχετικά μικρές πόλεις. Δεν έχουμε τεράστιες μητροπόλεις, τόσες πολλές και ίσως αυτό είναι καλό. Έχουμε 50 πόλεις όμως ε, των οποίων ο πληθυσμός ξεπερνά το 1 εκατομμύριο κατοίκους. Όμως το 75% των Ευρωπαίων πολιτών ζουν σε πόλεις κάτω του 1 εκατομμυρίου κατοίκων, ε, δηλαδή σε αστικά κέντρα ε, μικρομεσαία. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η οικονομική ανάπτυξη, το οποίο ουσιαστικά προϋποθέτει τις χρήσεις γης. Έχουμε 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα αστικής γης ή τεχνητής γης στην Ευρώπη, ενώ αρκετά τετραγωνικά χιλιόμετρα καλύπτονται κάθε χρόνο από τις πόλεις μας για λόγους οικιστικούς, για λόγους στέγασης και άλλους. Επομένως χάνουμε αρωτρέα γη, αρρώσιμη έκταση και αυξάνεται και το δίκτυο αποχέτευσης. Είναι δύσκολο να ανακτήσουμε εκτάσεις. Έχουμε διάφορες χρήσεις γης και διάφορες μορφές της που δεν είναι καθόλου βιώσιμες. Και όλα αυτά τα θέματα πρέπει μια ατζέντα για το άστι να τα χειριστεί και να τα αντιμετωπίσει. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για τη Στοκχόλμη. Μια πυκνοκατοικημένη πόλη, τη βλέπετε εδώ. Έχουμε μακρά παράδοση, παράδοση βιώσιμης χρήσης γης. Ήταν η πρώτη πράσινη πρωτεύουσα το 2010. Έχουμε μια πόλη συμπυκνωμένη δίκαιη για τους πολίτες, υπάρχει εγκύτητα, η κοινωνική διάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και να σας δώσω πέντε παραδείγματα για το πώς το κάνουμε, προσπαθώντας να εμπνεύσω και άλλες πόλεις. Εδώ βλέπετε πώς αντιμετωπίζουμε μια ε, πυκνή πόλη και την εγκύτητα στις δημόσιες μεταφορές. Έχουμε ε, δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσουμε να καταστήσουμε εφικτή αυτού του είδους την εξέλιξη. Είναι στα αριστερά το 2010 και στα δεξιά το 2020 που θέλουμε να φτάσουμε. Είναι εξαιρετικά δαπανηρό πράγματι για τους πολίτες, αλλά το 2020 θα ε, έχουμε αποτελέσματα. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί ε, η ανάκτηση των χρήσεων της γης. Βέβαια πολλές πόλεις δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Έχουμε την απορρίπανση και την ανάπτυξη τύπου Brownfield. Βλέπετε από το 1996 μέχρι το 2010. Το τρίτο είναι να, οι πράσινες, οι χώροι πρασίνου να παραμείνουν πράσινοι. Να προσπαθήσετε γι' αυτό. Βλέπετε τα νούμερα από το 98 μέχρι το 2009. Χάσαμε το 2% το χώρων πρασίνου ενώ ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 15%. Μπορεί να γίνουν τόσο μικρές απώλειες αλλά ε, χρειάζεται πολιτική βούληση. Το σημαντικό είναι να δημιουργηθούν συνέργειες για την προσαρμογή στην εξέλιξη των κλιματικών συνθήκων, για την προστασία των οικοσυστημάτων, ε, για να έχουμε σωστά συστήματα υπηρεσιών σε θέματα χώρο ταξίας και πόλεοδομίας δεν μιλούμε για χρήση γης μόνο για λόγους χτισήματος και κατασκευών, αλλά και για χρήση γης προκειμένου οι πόλεις να γίνουν πράσινες και να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. Εδώ έχουμε μικτές χρήσεις και μικτές ε, δομές και υποδομές. Δεξιά ένας μεγάλος δρόμος, μια μεγάλη λεωφόρος, η οποία μπορεί να αλλάξει και να πάρει τη μορφή που βλέπετε κάτω στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να γίνει αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε πολλούς περιορισμούς και ειδικότερα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα και για τα επίπεδα ηχορύπανσης. Το βασικό λοιπόν μήνυμα από τη Στοκχόλμη για τις χρήσεις γης είναι ότι απαιτείται σαφής πολιτικός σχεδιασμός, σαφής πολιτική άποψη και μακροπρόθεσμη δέσμευση. Αυτά τα δουλέψαμε στη Στοκχόλμη και ήταν αποτελεσματικά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα της ιδιοκτησίας της γης και έτσι ε, μπορεί κανείς να κάνει τα δέοντα για να πληρώσει και να χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα έργα και τα project. Η Ευρώπη έχει ρόλο να διαδραματίσει ως προς το πεδίο αρμοδιοτήτων. Μια εξελιγμένη μορφή διακυβέρνησης είναι απαραίτητη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όμως το να υπάρχουν σωστές μελέτες και καλή τεκμηρίωση και καλή παρακολούθηση στη συνέχεια της εφαρμογής και της εξέλιξης των έργων είναι εξαιρετικά σημαντικό θα έλεγα και θα το υπογραμμίσω ξανά και ξανά ότι προφανώς οι πόλεις πρέπει να εμπλακούν οι εκπρόσωποι τους σε οποιαδήποτε εργασία και προφανώς οι πόλεις θα πρέπει να χρηματοδοτούν όλα αυτά τα έργα καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να έχουμε μια οπτική γωνία όσο το δυνατόν πιο ε, ευρεία ε, γίνεται και να περιλάβουμε και την άποψη των μεγάλων μητροπόλεων και όχι μόνο την οπτική γωνία των πόλεων. Τώρα θα ήθελα να σας δείξω τρεις διαφάνειες για τους τρεις πυλώνες. Πρώτον, καλύτερη νομοθεσία. Γιατί η Στοκχόλμη είναι πολύ σημαντική αρχή της επικουρικότητας ως προς τις χρήσεις γης. Πράγματι, χρειαζόμαστε νομοθεσία και ευρωπαϊκή διάσταση στην νομοθεσία τη εθνική όμως, οι εμπειρογνώμονες σε κάθε πόλη, οι ειδικοί, θα πρέπει να αξιοποιούνται. Πρώτος πυλώνας λοιπόν καλύτερη νομοθεσία. Δεύτερος, χρηματοδότηση. Συμφωνώ και με τον Μάικλ. Ε, η χρηματοδότηση είναι που έχει τεράστιο αντίκτυπο στις πόλεις. Μια ε, καλή γη, μια έκταση σωστή πρέπει να αμυφθεί, να ανταμυφθεί αν θέλετε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να μην ξεχνούμε το, την πράσινη διάσταση των χρήσεων γης και ειδικότερα των αστικών οικοσυστημάτων. Και πρέπει να υπάρξει συνδυασμός με τις λύσεις για τις έξυπνες πόλεις, έτσι ώστε να διατηρηθεί η γη και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Τέλος, είναι απαραίτητη η μάθηση, οι ανταλλαγές απόψεων, εμπειριών, και να πλησιάσουμε τον πολίτη. Να, ειδικότερα όταν γίνεται λόγος για ισότητα μεταξύ διαφορών κοινωνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών για παράδειγμα. Πρέπει να προσεγγίσουμε τον πολίτη κάθε φορά που μιλούμε ή προωθούμε την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, ε, το άστι, για την αστική διάσταση ανακάλυψα ότι δεν γίνεται σωστή παρακολούθηση των χρήσεων υγιής στην Ευρώπη. Και είναι ένα μήνυμα που πρέπει να διαδοθεί. Χρειαζόμαστε καλύτερα νούμερα, πιο στέρεα, πιο αξιόπιστα στοιχεία για να χαράξουμε και πιο αξιόπιστη πολιτική. Και τέλος, μπορώ να σας πω ότι τα δίκτυα τα εφιστάμενα στην Ευρώπη πρέπει να αξιοποιηθούν για τα παραδοτέα ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ατζέντας για το άστι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, κάποιες προκλητικές, με πολλές πληροφορίες. Τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για ερωταπαντήσεις και συζήτηση. Δύο μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν στήσει το λόγο, αλλά θα ήθελα να ε, δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κατανέο, ο οποίος θα δώσει το λόγο στα μέλη της ΚΟΤΕΡ. Ο κύριος Πετερόσφαλτ έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις. Εγώ ασχολούμαι με το θέμα αυτό από το 1998 και έχω κάποια σχόλια για το πρόγραμμα της Βιέννης. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ε, πολλά υποσχόμενο. Θα ήθελα να πω όμως ότι πολλές φορές τα πράγματα είναι διαφορετικά στις πόλεις των νέων κρατών μελών, διότι οι πόλεις βρίσκονται σε στάδιο αλλαγής και εξέλιξης. Γι' αυτό πολλές φορές ο τομέας, για παράδειγμα, των μεταφορών έχει άλλες απαιτήσει. Είναι ένας τομέας που αλλάζει και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λύσεις της Βιέννης για αυτές τις πόλεις. Σε σχέση με τη χρήση του αστικού θεματολογίου στα επιχειρησιακά προγράμματα των πόλεων. Να σας πω ότι εξαρτάται από τα οικονομικά της κάθε πόλης και διαφορετικές δυνατότητες υπάρχουν σε κάθε πόλη και πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθεί αυτό στον σχεδιασμό. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τους πόρους της κάθε πόλης και από πού αυτοί προέρχονται. Κάποιοι προέρχονται μέσω της φορολογίας, κάποιοι μέσω των ε, μέσω της κυβέρνησης λοιπά. Το αστικό θεματολόγιο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα, διότι δεν θα εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη το σύστημα αυτό με τον ίδιο τρόπο. Κάποιες άλλες χώρες έχουν χαμηλό ενδιαφέρον και πιστεύω πως η μεθοδολογία και η νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κομισιόν ε, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Περιμέναμε δύο χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος για προτάσεις και γι' αυτό λοιπόν έχω τις αμφιβολίες μου για το αν κάποιος ε, θα προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Για παράδειγμα αυτήν την ε, πιστοποίηση των ITI. Ε, τώρα, για τον κύριο Πάρκινσον, να πω ότι με χαροποίησε πάρα πολύ η παρουσίασή σας και πιστεύω πως αποτελεί πολύ καλή βάση για την προετοιμασία ε, για το 2020 και 2027. Εάν θέλουμε να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά, πρέπει να αρχίσουμε από τώρα, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το μέλλον. Πολύ φοβάμαι όμως ότι ε, ήρθε και η παρουσίαση του κύριου Πάρκινσον πολύ αργά. Δέκα χρόνια πριν θα μπορούσαμε να την είχαμε χρησιμοποιήσει και να καταφέρουμε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτριά μας, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για την αστική διάσταση και στην Βέστφαλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω πολύ και πολύ δυνατά γιατί είμαι άρρωστη. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική έκθεση και την εξαιρετική μελέτη που μας παρουσιάσατε. Πραγματικά βοηθάτε πάρα πολύ εμάς ε, τους ε, ευρωβουλευτές και τα μέλη της Κοτέρο. Γιάννα Όλμπριχτ και εγώ αρχίσαμε ήδη τις ε, συζητήσεις για τη νέα, για τη νέα περίοδο και προσπαθήσαμε να εξετάσουμε όλες τις ε, πτυχές. Όμως εσείς με την ε, μελέτη σας και με αυτό που μας είπατε μας βοηθάτε πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Περιμέναμε 20 ολόκληρα χρόνια και επιτέλους τώρα καταφέραμε να ψηφίσουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Ε, χρειάζεται αυτή τη στιγμή να επιταχύνουμε, διότι όπως ακούσαμε και στην παρουσίαση του αγαπητού συναδέλφου, το 70% των Ευρωπαίων ζει σε ε, πόλεις, σε αστικά κέντρα και είναι η κινητήριος ε, δύναμη της ανάπτυξης η πόλης. Χρειάζεται όμως να τονίσουμε ότι, όπως αναφέρεται και στη δική μας ε, έκθεση και στην δική σας, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις μικρότερες πόλεις, τα μικρότερα αστικά κέντρα. Ας μην επικεντρωνόμαστε μόνο στις μεγάλες, στις μεγαλοπόλεις, στις μητροπόλεις. Διότι φοβάμαι ότι στο τέλος θα έρθουν σε αντιπαράθεση οι πόλεις με την Ήπεθρο και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Γι' αυτό και στην έκθεση συμπεριλάβαμε κάποια στοιχεία που ε, τονίζουν την καλή ε, συνεργασία και τη σημασία που έχει αυτή. Χρειάζεται επίσης μεγάλη προσοχή στους ε, υπεύθυνους, στους αρμόδιους, στους επικεφαλείς. Υπάρχει ένας αυτή τη στιγμή ε, υπάλληλο Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με τον συντονισμό. Δεν είναι αρκετό αυτό. Ο συντονισμός πρέπει να γίνεται σε περισσότερα επίπεδα για να είναι αποτελεσματικότερος. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία ε, βρίσκονται στην έκθεσή μας, για παράδειγμα το σύμφωνο του Άμστερνταμ και η αρχή των ε, εταιρικών σχέσεων. Όπως αναφέρατε και οι τρεις σας, υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό και όπως είπατε πρέπει όλοι οι φορείς να ε, συμπεριληφθούν. Διότι χωρίς ε, τη συμμετοχή τους δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς την οικονομική στήριξη όλων των φορέων δεν μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις λοιπόν τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως αναφέρατε η δημογραφική αλλαγή είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση αλλά και το στεγαστικό ε, ζήτημα. Χρειάζεται περισσότερη ε, κοινωνική στέγαση, κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό ζήτημα. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη γνώμη μας και η πολυμορφία των πόλεων. Έχοντας πει όλα αυτά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμότατα, διότι βοηθήσατε πάρα πολύ στο δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Δύσκολο, αλλά όχι εκατόρθωτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντάμοβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς όλους για τις παρουσιάσεις σας. Θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Έρμαν, με αυτά που μας είπε. Ήταν πολύ θαραλέα παρουσίαση. Όπως είπε και ο κύριος Έρμαν λοιπόν, αυτά τα έργα αφορούν κυρίως τις μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν όμως και ε, οι μικρότερες, οι μεσαίου μεγέθους πόλεις, τις οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε. η καινοτομία, και... η είναι χαρακτηριστικό των πόλεων. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη οικονομική ε, ανάπτυξη στις πόλεις και η οικονομική διάσταση μας λείπει από, ε, τις, ε, από το αστικό θεματολόγιο και πρέπει λοιπόν να συνδυαστεί. Εάν η Ευρώπη θέλει να συναγωνιστεί και να ανταγωνιστεί τις άλλες υπήρους πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτήν την πλατφόρμα για τις Μητροπόλεις. Ξέρουμε πως αστικοποιείται ο κόσμος και οι πόλεις ολένα και μεγαλώνουν. Δεν θέλω βέβαια η έκθεση να προσπαθήσει να ευχαριστήσει όλους, αλλά το αστικό θεματολόγιο πρέπει να ε, αντικατοπτρίζει τις ε, δικές μας ιδέες για την πολιτική και το αστικό θεματολόγιο στην Ευρώπη. Πιστεύω πως ο συνάδελφος από την Σουηδία είχε απόλυτο δίκιο. Οι πόλεις χαρακτηρίζονται από πολυμορφία. Υπάρχουν και διαφορετικού μεγέθους πόλεις. Κάποιες πόλεις μερικών χιλιάδων κατοίκων και κάποιες μεγάλου πόλεις εκατομμυρίων. Δεν μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μία λύση που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά να καταλάβουμε τις ιδιαιτερότητες της έννοιας πόλη και πιστεύω πως χρειάζεται γι' αυτό να δημιουργηθούν κάποια κριτήρια που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε περισσότερο το χαρακτήρα μιας πόλης. Τι είναι μια πόλη λοιπόν. Χρειάζεται να βρούμε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Για παράδειγμα, ένα από τα κριτήρια θα μπορούσε να είναι ο πληθυσμός. Και κάτι άλλο. Στη σελίδα 27 του αστικού θεματολογίου, βλέπουμε τα διάφορα επιμέρους θέματα και βλέπουμε μία πολυμορφία, από την οποία όμως λείπει ο πολιτισμός. Και είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυσή της χωρίς το στοιχείο του πολιτισμού. Χρειάζεται λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι οι πόλεις μας έχουν και δημογραφική κοινωνικά ζητήματα και προκλήσεις. Ε, γυράσκει ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα. Και επίσης οι πόλεις απαιτούν την συμμετοχή. Οι πόλεις έχουν ανοιχτό χαρακτήρα. Οι πόλεις πρέπει να δημιουργούν ένα αίσθημα οικειότητας και ε, ασφάλειας τους κατοίκους τους. Πρέπει λοιπόν να είναι ανοιχτές όχι προς τους ίδιους τους κατοίκους αλλά και προς τα έξω. Αυτόν λοιπόν τον ανοιχτό χαρακτήρα πρέπει να τον ενισχύσουμε διότι είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει περήφανους. Εμεί ευχαριστούμε τώρα το λόγο ο κύριο ο οποίο είναι μέλος του Περιφερειών αλλά επίση προεδρεύει στο Intergroup ε, για το Urban. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι από εμάς εδώ συμμετέχουν το Intergroup που είπατε αλλά και στην ε, ε, Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής παρατηρήσεις και ερωτήσεις πρώτα για να δούμε τι θέμα έχουμε στη σημερινή συνάντηση. Το θέμα μας είναι το σύμφωνο του Άμστερνταμ συνέπεια του θεματολογίου. Αυτό συζητούμε τώρα. Και το Μάιο στο θα εγκριθεί αυτό το σύμφωνο. Επομένως για αυτό και τον λόγο έγγραφο ε, δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Μία παρατήρηση τώρα. Εγώ είμαι εισηγητής για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού και του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και στην αναθεώρηση λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει πρόταση για το νέο ε, πολιτέ πλαίσιο πριν το τέλος του 2017. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει μια πρόταση δομημένη για το MFF και επίσης τι νέε πολιτικές που θα καλύψει αυτό το πολίτες πλαίσιο και επίσης προτάσει για την πολιτική συνοχής προ του τέλους του 2017. Το δε σύμφωνο του Άμστερνταμ εισάγει αυτές τις εταιρικέ σχέσεις που θα κρατήσουν τριετία. Δηλαδή 16-17 έως το 18 Επομένω, θα ολοκληρωθούν αυτέ οι εταιρικέ σχέσει αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει τη νέα τη πρόταση. Άρα θα πρέπει αυτό να μην το ξεχνούμε. Δεν υπάρχει χρόνο. Άρα θα πρέπει να δούμε ε, τα επιτεύγματα τη εταιρική σχέση στην εξέλιξη. Γιατί έχουμε τι πόλει, τα κρατή-μέλη, τους εμπειρογνώμονε. Δεν υπάρχει χρόνο να περιμένουμε μέχρι το τέλο Τότε θα είναι πολύ αργά. Μετά θα πάμε για 2027. Αυτό ήθελα να σας πω. Είναι παρατήρηση που δεν θα πρέπει να την ξεχνούμε. Είναι οι δυναμικές, η δυναμική. Κάτι άλλο τώρα. Ίσως μετά το δεύτερο τμήμα. Το, το ποιος θα το κάνει, ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω αυτό θα το ε, εξηγήσουν γιατί θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια γιατί ξέρουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία αφορά ή δεν αφορά το νορ πάντε καλέ αλλά τελικά πόσοι θα ασχοληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πόσοι θα είναι αρμόδιοι. Γιατί είπαμε, ο πύχη των φιλοδοξιών είναι πολύ ψηλά, να είμαστε συγκεκριμένοι. Τι γίνεται, πώ θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Μάικλ, πάρα πολύ προκλητικά τα, τα είπε σήμερα. Αλλά τώρα να είμαι και εγώ προκλητικός να σε προκαλέσω να μας πεις κάτι ξεκάθαρα πρώτα-πρώτα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οποίο είπες είναι ότι θα πρέπει συνέχεια να δίνουμε τη μάχη μας και ότι αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι το θεματολόγιο αλλά χρειάζεται μια πολιτική. Είναι ξεκάθαρο επίσης το σύμφωνο του Άμστερνταμ αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πόλεις και όχι το θεματολόγιο είτε μας αρέσει είτε όχι. Εάν κατάλαβα ότι λες επομένω συμφωνούμε 100%. Τα είπαμε και στην έκθεσή μας. Ή θα έχουμε ε, ε, αυτού είδου το εγχείρημα είτε θα έχουμε την πολιτική. Οπότε δεν χρειάζεται το εγχείρημα. Αλλά τι θα γίνει με την περιφερειακή πολιτική. Η πολιτική για τις πόλεις είναι τμήμα της περιφερειακής πολιτικής. Είναι άλλη πολιτική που ασκείται παράλληλα με την περιφερειακή. Να η πρόκλησή μου. Να απαντήσει γιατί αν δεν απαντήσει τότε θα είμαστε στο μετέχμιο. Θα είμαστε σε κάποια συζήτηση πολύ τεχνητή και θα έχουμε την τύχη του Urban εν προκειμένου επίσης. Άρα, τι γίνεται με αυτές τις δύο πολιτικές. Είναι η μία αντιπαρατηθέμενη στην άλλη πρόεδρος. Ο χρόνος κυλά. Και έχουμε και ένα δεύτερο τμήμα στην ε, συζήτηση της επόμενης εισηγήσεις. Τώρα έχουμε τρία μέλη της Επιτροπής Περιφερειών που ζητήσει το λόγο, συμπεριλαμβανομένων και των δύο συγκητών, Νταγκελόπερ και Φερχάκεν, αλλά Εάν έχουμε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα, να σας δώσω το λόγο. Αν επομένω πρέπει να ακούσουμε το ερώτημα τώρα. Από την άλλη μεριά όμως, αν πρόκειται για γενικότερες παρατηρήσεις, τότε καλύτερα να κάνουμε πρώτα τις εισηγήσεις και στη συνέχεια να λάβουν τον λόγο τα μέλη των ε, περιφερειών και βεβαίω τη Επιτροπή Περιφερειακή Πολιτική για το δεύτερο και τελευταίο τμήμα τη ε, συζήτηση πριν τι καταληκτικέ παρατηρήσει. Συμφωνείτε? Υπάρχει κάποιο ερώτημα. Όχι. Ναι, ναι. Λέει συμπρόεδρος. Ναι, μα υπευλήθηκε το ερώτημα του κυρίου Όλμπριχ προς τον κύριο Πάρκινσον. Μπορείτε να απαντήσετε. Δεν ήταν αρκετά προκλητικός για να προκαλέσει την απάντηση. Αυτός μέση εδώ στις Βρυξέλλες για να Σα πω αυτό που σα λέω, για λογαριασμό του. Λέω κ. Πάρκινσον, να σα τα πω έξω από τα βράδια. Τώρα δεν έχω καμία δεσμεύση. Λέω ό,τι θέλω. Να τι πάνε πει πανεπιστημιακό, διότι έχω μπουχτίσει να έρχομαι εδώ επί 25 χρόνια στι Βρυξέλλε και να συζητάμε για πράγματα να μην γίνεται τίποτα. Και συμφωνώ 100% γιατί νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ε, λέμε ότι έχουμε θεματολόγιο και όλα να απονευρώνονται, όμως θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική και πολιτική για τις πόλεις. Να είναι πολύ πολυδιάστατη, ε, πολύπλοκη και όπως είπε ο συνάδελφος θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είδους Ευρώπη θέλουμε, τι ρόλο θέλουμε να παίζουν οι πόλεις μας, τι έχουμε πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε, τι θα κάνουν τα κρατή μέλη, τι θα κάνουν γενικές ε, διευθύνσεις, τι θα κάνουν οι περιφέρειες, να είμαστε πολύ περισσότερο συγκεκριμένοι. Έχει δίκιο ο Άλμπρεχτ. Θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες υλοποίησης. Τα διάβασα και είπα ότι να είναι το σύμβολο του Άμστερνταμ. Πάει και πάλι λόγια, λόγια. Ποιος θα τα υλοποίησε. Όχι, δεν θα συνέχιζα την περιφερειακή πολιτική. Θα το ονόμαζα πολιτική για τις πόλεις. Αυτό θα είναι κίνητρο για τα κρατημέλη. Και άλλωστε ο διαχωρισμός περιφέρειας από την πόλη είναι κάτι το απαρχαιωμένο. Ας αποφασίσουμε σε ποιο επίπεδο κάνουμε ποια κίνηση. Το είπε πριν και ο συνάδελφος ή η συνάδελφος. Χρειάζεται μια ξεκάθαρη πολιτική για τις περιφέρειες των πόλεων και για τις περιφέρειες σκέτο. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε ούτε να δούμε τις ευκαιρίες ούτε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να μετακινήσουμε το κέντρο προσοχής και αν θεωρήσουμε ότι τώρα πάμε στην περιφερειακή πολιτική για τις πόλεις δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πρέπει να πούμε τόσο για, τους, το τόσο για τις πόλεις ανάλογα με το ποσοστό του ΑΕΠ να πώς απαντώ στην πρόκληση ε, ευχαριστώ λέει πρόεδρος Άρα βλέπουμε τώρα συζήτηση πάει να γίνει συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και για τις πόλεις όμως. Οπότε τώρα ας συνεχίσουμε με τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων μας. Έχουμε τώρα την ε, κυρία Γελένα Ρίκοφ που προέρχεται από την Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο γραφείο του Ζάγκρεβ για προγράμματα και έργα. Σε με την ε, φτώχεια, με προσβασιμότητα, σε στέγαση, σε σχέση με τις ε, δημοτικές αρχές της πόλης. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω υπό την οπτική γωνία των, της τοπικής αυτοδιοίκησης πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις για προσβάσιμη στέγαση και ελπίζω να αναδείξω πως οι ΙΟΤΑ μπορούν να συμβάλλουν ε, στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Βλέπετε στην οθόνη ορισμένα γεγονότα πολύ εύγλωτα θα έλεγα, τα γνωρίζετε ήδη. Το 70% του πληθυσμού στην Ευρώπη ζει σε αστικά κέντρα και οι περισσότερες ε, πολιτικές που εφαρμόζονται επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων στις αστικές περιοχές. Όμως δεν έχουμε ατζέντα για το άστι και ε, συμμετοχή αυτή στη διαβούλευση. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί η διαδικασία της επιτροπολογίας έτσι ώστε να εμπλέκεται με συστηματικό τρόπο κάθε οτά στην ε, κατανομή των κονδυλίων, στη χρηματοδότηση και στη χάραξη των πολιτικών. Είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί επανειλημμένως και φάνηκε και με την διετή συνεργασία της Επιτροπής Ρέτζη και της Επιτροπής Κοτέρ, που υιοθέτησαν διάφορες πρωτοβουλίες και κατέληξαν στην έγκριση συγκεκριμένου κειμένου. Εάν δούμε όλα αυτά τα έγγραφα, ε, θα έλεγα ότι πολύ σωστά αρθρώνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις και οι πολίτες και το, η πρόκληση που είναι το να έχει κανείς πρόσβαση σε προσβάσιμη στέγαση, σε προσβάσιμη στέγη. Ωστόσο, Όλα αυτά τα αντιμετωπίζει καλύτερα η τοπική αυτοδιοίκηση, το τοπικό επίπεδο διαχείρισης και διακυβέρνησης που μπορεί να προτείνει λύσεις για τη σωστή διοχέτευση των πόρων και για τη δράση εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται η ανάληψη δράσης. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα θέματα ε, συνεχώς αλληλοκαλύπτονται, αλληλοεπικαλύπτονται και λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω της πρόσφατης μεταναστευτικής κρίσης. Όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεθεμένα μεταξύ τους. Δηλαδή το ότι η αστική φτώχεια επεκτείνεται και ότι η ανάπτυξη στέγασης που να ταιριάζει ε, στις πόλεις είναι κάτι που είναι επιτεκτική ανάγκη, ε, όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία ε, αλληλοσημαίονται άρρηκτα. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι μεγάλο και σοβαρό, αλλά για να μπορέσουν οι πολίτες να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες που είναι ένα σπίτι, διατροφή, εκπαίδευση, ε, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ε, τις οποίες καλούνται οι πόλεις να παράσχουν. Όλα αυτά τα νούμερα είναι πολύ εύκολα τα που βλέπετε στην οθόνη. Ως προς τη στέγαση, αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη είναι ότι δεν υπάρχει μία ενιαία πολιτική, ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Τεράστιες είναι οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για κοινωνική στέγαση ενώ μειώνονται τα οικιστικά έργα για κοινωνική στέγαση ή εργατικές κατοικίες από τις πόλεις. Έχουμε απώλεια θέσεων απασχόλησης και απώλεια κατοικίας για πολλούς ανθρώπους. Αυτό επίσης από την άλλη λόγω της λιτότητας μειώνεται ο προϋπολογισμός των δήμων των πόλεων, λιτότητα που εφαρμόζουν οι εθνικές κυβερνήσεις και έχουμε και τους κανόνες για την κρατική ενίσχυση όταν μιλούμε για υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, οι οποίοι κανόνες δεν βοηθούν καθόλου, γιατί είναι πολύ ε, περιορισμένη η πρόσβαση, ανοίγεται αν θέλετε η κάνουλα μόνο στις πολύ μειονεκτικές και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όλα αυτά καθιστούν δύσκολο να υποστηρίξουμε το εφιστάμενο μοντέλο ε, ε, κοινωνικής στέγασης. Σε αυτό το πίνακα βλέπετε το πρόβλημα και το μέγεθος του, το πρόβλημα στέγασης. Και αυτό δεν καταγράφεται, ξέρετε, συχνά. Μιλούμε για νέους ενήλικες που ζουν με τους γονείς τους. Μέσα στα 34. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, έχουμε περιοχές όπου το 50% των νέων ενηλίκων μέχρι 34 ετών ζουν με τους γονείς τους. Δεν νομίζω ότι όλοι το επιθυμούν από αυτούς. Απλά δεν έχουν τα οικονομικά μέσα, δεν έχουν πρόσβαση σε ένα σπίτι το οποίο να μπορούν να πληρώσουν ε, σε μια κατοικία. Πώς αντιμετωπίζουν λοιπόν οι πόλεις το θέμα αυτό. Αντιμετωπίζουμε συνεχώς επιπρόσθετα αιτήματα στήριξης από τους πολίτες μας. Δεν υπάρχει ένα μόνο ενιαίο μοντέλο. Έχουμε τις δυτικές χώρες που έχουν μακρά παράδοση ε, κοινωνικής στέγασης, κοινωνικών κατοικιών, π.χ. στην πόλη της Βιέννης, η οποία ξεκίνησε να χτίζει τέτοια σπίτια από το 1920, ενώ σήμερα το 25% των κατοικιών στη Βιέννη ανήκει στο Δήμο και έχουμε από την άλλη τις μετακομμουνιστικές χώρες ή τις ανατολικές χώρες με άλλα λόγια, όπου πριν από τη μετάβαση όλα άνοικαν στο κράτος, ήταν κοινωνική κατοικία όλων. Μετά τις ιδιωτικοποίησεις όμως έχουμε ένα τεράστιο κενό για τους ε, φτωχούς πολίτες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην άνοδο των τιμών ε, της ιδιοκτησίας που πέρασε σε, ε, στα χέρια ιδιωτών. Αυτό ισχύει για παράδειγμα ε, στην πόλη του Ζάγκρεμπ. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα κατοικιών, κατασκευής και κατοικιών πριν από 15 χρόνια. 5.000 διαμερίσματα χτίστηκαν και θα έρθουν και περισσότερα. Όμως, θελήσαμε να έχουμε και κοινωνικές υποδομές, γιατί το να χτίσουμε κατοικίες δεν λύνει, πρόβλημα, ε, δεν λύνει το πρόβλημα σε κάθε γειτονιά, από μόνο του. δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφοριών, πολιτικών, εμπειριών, βιωμάτων από τις διάφορες πόλεις. Νομίζουμε ότι μια ατζέντα για το άστι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το απαιτήσει αυτό. Και σε αυτό αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όχι για όλες τις χώρες αλλά σίγουρα για τις ανατολικές χώρες, τις χώρες του Νότου συμπεριλαμβανομένες της Ιταλίας και της Κροατίας. Είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δηλαδή έλλειψη προσβάσιμης κατοικίας είναι ένα φαινόμενο το οποίο οδηγεί ε, σε ε, αυθαίρετες κατασκευές παράνομες παράτυπες. Στην Κροατία έχουμε μια διαδικασία νομιμοποίησης αυτών των αυθαίρετων κατοικιών και επειδή δεν έχει γίνει χωροτοξική και πολεοδομική μελέτη, τα αυθέρατα δεν έχουν πρόσβαση σε δέκο. Και αυτό δημιουργεί ε, προβλήματα υγιεινής, ασφάλειας και τελικά θα κάνει όλες αυτές τις περιοχές να γκέτοποιούνται. Εδώ βλέπετε λοιπόν πως το πρόβλημα της φτώχειας αλληλοδικαλύπτεται με το πρόβλημα ε, της έλλειψης επαρκούς κοινωνικής στέγασης. Τώρα, ως προς τη φτώχεια έχουμε ακόμα πιο σχετικά νούμερα και δεδομένα. Πέρα από το γεγονός ότι όχι μόνο δεν μειώσαμε τη φτώχεια στην Ευρώπη, αντιθέτως έχει αυξηθεί η φτώχεια, έχει περιλάβει α, άλλους 7 εκατομμύρια ανθρώπους, 5,1 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άστεγοι, πάρα πολλοί δεν μπορούν να πληρώσουν θέρμανση, και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού κινδυνεύει με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Όλα αυτά συμβαίνουν τα τελευταία 5 ή 10 χρόνια, καλύτερα 5 μάλλον χρόνια, λόγω των διαφόρων πολιτικών που υιοθετήθηκαν για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα των χωρών. Και λόγω των οικονομικών πολιτικών που δημιουργήθηκαν, αυτές γέννησαν ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο κατά τη είναι μεγαλύτερο και έχει πολλαπλασιαστικό συντελεστή. Η ατζέντα για το άστι είναι μια πλατφόρμα έτσι ώστε να αναλύσουμε τις πολιτικές και να βεβαιωθούμε ότι προσπαθώντας να κάνουμε ένα καλό δεν ε, χαλάμε αν θέλετε το διπλανό του. Τώρα, εξετάζοντας τα έγγραφα, τις αιτίες, τα αποτελέσματα της φτώχειας στο άστι, βλέπουμε ότι το 2013 ε, ο αρμόδιο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπή αναγνώρισε ότι η φτώχεια είναι υψηλότερη στις πόλεις παρά στην Ήπεθρο ή στις μικρότερες κομοπόλεις. Και είναι υψηλότερη η φτώχεια στις πιο ανεπτυγμένες χώρες κιόλα. Και αυτό νομίζω ότι πραγματικά χτυπά το καμπανάκι του συνέγερμου, διότι είναι προφανές ότι ακόμα και πιο προηγμένες δυτικές χώρες έχουν μεγάλες μετροπολιτικές εκτάσεις, όπου είναι τεράστιο το πρόβλημα και δύσκολα αντιμετωπίζουν αυτές οι μετροπολιτικές περιοχές το θέμα της φτώχειας. Εμείς στην πόλη του Ζάγκρεπ ε, γινόμαστε συνεχώς μάρτυρες της όξυνσης του προβλήματος της φτώχειας στο άστι καθημερινά και ανακαλύπτουμε νέες μορφές φτώχειας, για παράδειγμα παιδική φτώχεια. Είναι συχνά κρυφή και μη καταγεγραμμένη, γιατί τα παιδιά πάνε στο σχολείο θα μπορούσαν να ανήκουν σε κανονικές οικογένειες αν θέλετε, αλλά τελικά να υστερούν σε επίπεδο υγείας, ε, φροντίδας, ή να μην ε, έχουν τραφεί επαρκώς. Στην Κροατία πέρσι για πρώτη φορά καταγράψαμε ότι υπήρχαν παιδιά που δεν μπορούσαν να αναλάβουν ε, τα οικονομικά οι γονείς τους τα έξοδα του γεύματος. Οι δάσκαλοι ενημέρωσαν τα μίντια, τα μίντια της πόλης και η πόλη στην κεντρική κυβέρνηση. Ωστόσο όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει ένας νέος τρόπος ανείχνευσης, εντοπισμού και μέτρησης των νέων μορφών φτώχειας. Ε, φτώχεια ε, στη στέγαση, στην υγεία, στην παιδική φτώχεια. Θα πρέπει να έχουμε μια νέα έννοια, μια νέα αντίληψη κοινωνικής φροντίδας, γιατί αυτές οι νέες μορφές φτώχειας είναι εξαιρετικά σημαντικές ε, ως οικονομικοί δείκτες. Μας επιτρέπουν να ε, αντιληφθούμε καλύτερα τις πολιτικές που θα χαράξουμε για την κατανομή των κονδυλίων και των προγραμμάτων των χρηματοδοτικών. Εδώ είναι ένας άλλος πίνακας που δημοσιεύω διότι δείχνει το ποσοστό των ανθρώπων με εισόδημα κάτω του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος και από τη μία και ε, του κόστου στέγασης από την άλλη. Δεν θα ήταν εξαιρετικά ανησυχητικό αυτός ο πίνακας εάν το κόστος στέγασης δεν ήταν τόσο μεγάλο. Εάν είναι τόσο μεγάλο το κόστος στέγασης είναι πολύ λίγα τα χρήματα που μένουν στον οικοκυριό για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των τροφίμων, ε, της εκπαίδευσης ε, και βεβαίως του πολιτισμού των αθλημάτων που είναι και αυτά απαραίτητα. Τα νούμερα λοιπόν είναι ανησυχητικά και εύγλωτα. Μιλάνε από μόνα τους και παίρνουν το μήνυμα πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε εμείς. Θα έλεγα ότι εμείς στις, ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση είμαστε στην εμπροστοφυλακή. Προσπαθούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες των πολιτών καθημερινά επί τόπου, σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, εάν γίνει έξωση σε μια οικογένεια γιατί δεν μπόρεσε να πληρώσει το δάνειο για το σπίτι, δεν θα πάει η, υποθήκη στο η οικογένεια στο Υπουργείο ούτε στην αρμόδια επιτροπή, θα χτυπήσει η οικογένεια την πόρτα του Δήμου και πρέπει εμείς να δώσουμε επίγον καταφύγιο και πρέπει να δούμε και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τι θα γίνει με αυτές τις οικογένειες. Εμείς λοιπόν δίνουμε βοήθεια, τους βοηθάμε να ξανασταθούν στα πόδια τους, ε, να βρουν δουλειά, ε, τους δίνουμε διάφορες μορφές βοήθειας. Αυτά κάνουμε καθημερινά. Και παρόλο που η πόλη του Ζάγκρεπ άνω του 30% του ετήσιου προϋπολογισμού της, ε, ε, το δίνει η πόλη του Ζάγκρεμπ σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε τη δικαιοδοσία μιας κοινότητας, δηλαδή ε, του Δήμου. Είμαστε υπεύθυνοι και για τις, τους συνταξιούχους και για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και για τα νηπιαγωγεία, τους παιδικούς σταθμούς, τα δημοτικά, ε, μεταξύ άλλων σχολεία. Δηλαδή έχουμε τεράστια εμπειρία, εκτιθέμεθα σε όλες τις ανάγκες, βλέπουμε ανα πάσα στιγμή τι είδους στήριξη χρειάζεται, σε ποια μορφή και πότε και πού Επομένως έχουμε πολύ πιο γρήγορο feedback, πολύ πιο γρήγορη ανατροφοδότηση για το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Είμαστε ε, σε καλύτερη θέση και μπορούμε να προτείνουμε καλύτερα στην Εθνική Κεντρική Κυβέρνηση ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να προτείνουμε τι πρέπει να γίνει και μάλιστα αμέσως και όχι σε 20 χρόνια όπως είπαν άλλοι συνάδελφοι ότι συζητούνται τα θέματα αυτά. Να σα υπενθυμίσω, λέει η πρόεδρο, ότι πρέπει να συντομεύετε. Ε, μάλιστα κύριε Πρόεδρε, ε, ολοκληρώνω. Λέγοντα ότι Πράγματι οι πόλεις προσπαθούν να είναι καινοτόμε και να βρίσκουν λύσει και εμεί αυτό πράττουμε από την πόλη του Ζάγκρεπ. Ε, μπορώ να επιβεβαιώσω ξανά, ε, δεν είναι ότι θέλω να το επαναλάβω, είναι ότι θέλω και εγώ με τη σειρά μου να το υπογραμμίσω αυτό που είπαν οι προηγούμενοι εισάδελφοι που πήραν το λόγο προηγουμένω. Αυτό που λείπει είναι μια μονοαπευθυντική θηρίδα ε, ένα σημείο στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα συνομιλητής στον οποίο μπορούμε να εκμυστηρευτούμε τις ανησυχίες μας, να υποβάλουμε προτάσεις και μέσω αυτού να συμμετάσχουμε στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Περιμένουμε με αγωνία και με μεγάλη προσδοκία ε, να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωση της ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα αστικά κέντρα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ο κύριος Κατάνεο. Ε, σας ευχαριστώ να παρουσιάσω τον επόμενο ομιλητή, Ραμόν Σανναπούκα, ε, αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης διαπολιτισμικότητας στη Βαρκελόνη. Είναι, ε, συμμετέχει στη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο EuroCities και σήμερα θα μας μιλήσει για την πρόκληση της μετανάστευσης και των προσφύγων στην πόλη της Βαρκελόνης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. για την πρόσκληση να σας παρουσιάσουμε την άποψη της Βαρκελόνης για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών. Πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για μια νέα αστική πολιτική και ένα νέο αστικό θεματολόγιο. Και η προσφυγική κρίση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ε, το κάνουμε αυτό λαμβάνοντας υπόψη τις ε, αστικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Πρωτού αρχίσω, θα ήθελα να... Με συγχωρείτε, λέει ο μιλητής, κάποιο τεχνικό πρόβλημα προέκυψε. Θα αρχίσω λοιπόν με κάποιες εικασίες σχετικά με την ε, μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική στο τοπικό και κρατικό επίπεδο. Καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλες οι όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχουν εξαιτία τη μετανάστευση. Χωρίς μετανάστευση δεν θα υπήρχαν πόλεις. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η μετανάστευση είναι αμφίδρομη διαδικασία. Και οι μετανάστες αλλά και οι ντόπιοι συνεργάζονται. Είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και το συγκείμενο, όπω είπε και ο συνάδελφο από τη Σουηδία. Την ιστορία μια πόλη, την εθνική νομοθεσία, τον κοινωνικό ιστό, το πολιτικό σύστημα, τι πολιτικέ, το τι δηλαδή συνιστά μία πόλη και να αναγνωρίσουμε τις διαφορές στην κάθε περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες στην ένταξη μεταναστών και προσφύγων. Δεν υπάρχει μία νέα λύση και εδώ Είμαστε ανοιχτοί στην συζήτηση. Αργότερα θα εξετάσω κάποιες επιμέρους περιπτώσεις. Θα συνεχίσω όμως τώρα λέγοντας ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την πολιτική ένταξη ολιστικά. Όχι μόνο δηλαδή από οικονομική άποψη, από κοινωνική άποψη, αλλά συνολικά. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Η ασφάλεια, η ανάπτυξη, και οικονομία. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη εδώ ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκες. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι ουδέτεροι, έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία, διότι πρέπει να συζητήσουμε για τη στέγασή τους, για την ένταξή τους στο σύστημα υγείας, για, την, ε, για τις δραστηριότητες αναψυχής, για την απασχόλησή τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι η ένταξη είναι τοπική αρμοδιότητα. Είναι κάτι που συμβαίνει στη συγκεκριμένη πόλη, στη συγκεκριμένη γειτονιά. Και θα ήθελα εδώ να εξετάσω ορισμένους συμβιβασμούς που έχουμε κάνει. Για παράδειγμα, κρατική αρμοδιότητα ε, σε αντιπαράθεση με την τοπική αρμοδιότητα. Κρατική αρμοδιότητα έχει να κάνει με το ποιο μπαίνει στην Ευρώπη, ποια είναι η νομοθεσία που τους ε, καλύπτει, πώς αποκτά κάποιος πρόσβαση στην ε, διαδικασία απόκτησης ηθαγένειας. Υπηκότητας, με συγχωρείτε. Πρωτού λοιπόν αρχίσουμε να ε, συζητούμε την πολιτική συνοχή, πρέπει να δούμε πώς ε, γίνεται η διαδικασία ένταξης, με ποιον τρόπο συντελείται αυτό. Όπως είπα και προηγουμένως, όλα συνδέονται. Εάν το κράτος περιορίζει ε, τις ε, πολιτικές του, η ένταξη είναι πιο δύσκολη. Εάν το κράτος περιορίζει τις πολιτικές ε, επανένωσης με την οικογένεια, αυτό έχει επιπτώσει στην ποιότητα ζωής των μεταναστών μας. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μετανάστες και πρόσφυγες. Υπάρχει καταρχάς ο νομικός ορισμός των κρατών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Γενέβης. Αυτά τα κράτη έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν τους πρόσφυγες από όπου και αν προέρχονται. Ωστόσο, οι πολιτικές ένταξης προσφύγων και μεταναστών μακροπρόθεσμα είναι περίπου ίδιες. Υπάρχει νομική υποχρέωση από τα κράτη για να προστατεύουν τους πρόσφυγες, να τους δίνουν καταφύγιο και αυτό ισχύει και για τους ε, μετανάστες. Εδώ υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Ευρώπη. Η Βόρεια Ευρώπη ε, χαρακτηρίζεται από διάφορα προγράμματα αιτήσεων ε, ασύλου. Ένας πρόσφυγας πηγαίνει και ζητά άσυλο στην Βόρεια Ευρώπη. Στην Νότια Ευρώπη γίνεται το αντίστροφο. Υπάρχει νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται επαρκώς για το άσυλο και υπάρχουν πάρα πολλοί ε, μετανάστες, ε, νόμιμοι ή παράτυποι. Και οι δύο, και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι εξίσου σημαντικοί. Ωστόσο, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκει πολύ περισσότερους ε, πρόσφυγες, πολύ περισσότερους ανθρώπους που ζητούν άσυλο. Στην περίπτωση της Ισπανίας υπάρχουν πολλοί μετανάστες και ελάχιστοι πρόσφυγες. Στο βορρά, βορρά της Ευρώπης υπάρχει το ίδιο, πολλοί πρόσφυγες και λίγοι μετανάστες. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσουμε την ε, πραγματικότητα των παράτυπων και νόμιμων μεταναστευτικών ροών. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποιος ε, στον οποίο θα αρνηθεί η χορήγηση ασύλου θα παραμείνει στη χώρα ως παράτυπος μετανάστης. Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να βρει δουλειά, στέγη. Εμείς στη Βαρκελόνη συνεργαζόμαστε με όλους και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας σε όλους ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του κάθε ανθρώπου. Και κάτι, μία ερώτηση νομική. Τι θα γίνει στην Ευρώπη μετά την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου όλων αυτών των ε, προσφύγων. Μιλάμε για 300.000 ανθρώπους, οι οποίοι τι θα κάνουν, θα πάνε στη Συρία πίσω, όχι. Θα παραμείνουν στις πόλεις μας όσο παράτυποι μετανάστες και δεν θα απελαθούν. Θα προσπαθήσω τώρα να παρουσιάσω ορισμένα συνενετικά μέτρα. Εμείς συνεργαζόμαστε με διάφορες άλλες πόλεις από όλη την Ευρώπη, με συντηρητικούς ή προοδευτικούς δημάρχους και καταφέραμε να καταλήξουμε σε ορισμένους ε, συνεντικούς ε, συμβασμούς σε αυτό το δύσκολο θέμα. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τι έχουμε καταφέρει σε τοπικό επίπεδο. Ως ε, συνέχεια της έκθεσης μας, την οποία μπορείτε να βρείτε όλοι, καταλήξαμε στην συνένεση ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική ηγεσία. Οι δήμαρχοι της κάθε πόλης πρέπει να κάνουν πολιτικές δηλώσεις σχετικά με το σύστημα, σύστημα της ε, ένταξης. Δεν πρέπει να φοβούνται να συζητήσουν για το μεταναστευτικό, διότι είναι κάτι που αφορά τους πολίτες και είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Υπάρχει επίσης ανάγκη διοργανικής συνεργασίας στα διάφορα επίπεδα διοίκησης αυτό είναι ένα γεγονός που έχουμε αναγνωρίσει σε πολλές χώρες ε, που έχει καταρρεύσει το σύστημα διεκπαιρέως αιτήσεων ασύλου. Έχουμε δει την πραγματικότητα ότι πολλές χώρες ε, πρέπει να συνεργαστούν, να υπάρχει επικοινωνία σχετικά με το πώς θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία. Επίσης, κάτι εξίσου σημαντικό είναι η δημιουργία νέων πολιτικών. Αυτή η κουλτούρα υποδοχή στη, στα γερμανικά κουλτούρα πρέπει να στηρίζεται η εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής, πρέπει να εξηγήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ε, τους νόμους μας, την παράδοσή μας, το πώς λειτουργούμε. Πρέπει να διευκολύνουμε επίσης την πρόσβαση στην ε, υγεία και στην εκπαίδευση. Και την κοινωνική ένταξη. Ας δώσουμε λοιπόν πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους στις υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση. Είναι μια επένδυση η οποία θα αποβεί καρποφορά στο μέλλον. Οι δήμοι μας πρέπει να εργαστούν έτσι ώστε να φαίνεται η πολυμορφία της κάθε πόλης. Και σε αυτό θα βοηθήσει πολύ η πολιτική ένταξη. Τέλος, έχουμε κάποιες συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερου χαρακτήρα. Καταρχάς, οικονομικές, πολιτικές και περιφερειακές πολιτικές θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ε, να υπάρχει άμεση πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης και επίσης οι πόλεις έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ηγετικό ρόλο σε αυτές τις ε, πολιτικές. Χρειάζεται επίσης πρόσβαση και καλύτερη χρησιμοποίηση του ΑΜΙΦ, του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Στην Ισπανία έχουμε πρόβλημα ε, στην χρήση αυτού του ταμείου, δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Και γεγονός είναι ότι τον τελευταίο χρόνο στην Ισπανία <clears throat> δεν έχουμε μπορέσει να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια από αυτό το ταμείο. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο διαστάσεις, και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και οι δύο ομάδες πρέπει να υποφεληθούν από αυτό το Ταμείο. Επίσης, χρειάζεται καλύτερη προσοχή στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη μετανάστευση. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα πρέπει να ενταχθούν στη ζωή της ε, πόλης υποδοχής και πρέπει επίσης να σκεφτούμε το τι θα γίνει μετά, μετά την ένταξη αυτών των μετανάστων και προσφύγων στην Ευρώπη. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσουν οι πολιτικές μας και τι αποτέλεσμα θα έχουν. Και τέλος, κάτι πολιτικό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα της παράτυπης μετανάστευσης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν παράτυποι μετανάστες και με αυτό πρέπει να προχωρήσουμε. Τέλος, λογοδοσία και διαφάνεια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης είναι κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουν τα κράτη-μέλη. Η λογοδοσία για τα προηγούμενα προγράμματα και για τη χρηματοδότηση. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι έγινε τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ισπανία με τα διάφορα ταμεία ένταξη. Τι έγινε λοιπόν με τα προηγούμενα κονδύλια. Όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν τα κονδύλια, όμως σε ποιες χώρες είδαμε αποτελέσματα. Υπάρχει κάποια χώρα η οποία δεν χρησιμοποίησε το 100% των κονδυλίων. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε αυτά τα στοιχεία για να γίνει μια αξιολόγηση. Έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει το αστικό θεματολόγιο. Τέλος, θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα του τι κάνουμε εμείς στη Βαρκελόνη. Χρησιμοποιούμε ένα διαπολιτισμικό μοντέλο το οποίο δίνει έμφαση στην διαπολιτισμικότητα και την ισότητα. Το λέμε convivencia, συμβίωση. Έχουμε κάποια πολύ ε, καλά πιστεύω παραδείγματα κοινωνικής πολιτικής. Καταρχάς, συστήνουμε ε, κάθε άνθρωπος που φτάνει στην ε, πόλη μας να αφομοιώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε την ένταξη για όλους και τα αστικά μητρώα, το, τα παδρών είναι μια καινοτομία της ε, Βαρκελόνης, τα δημοτικά μητρώα, τα οποία ε, χρησιμοποιούμε ε, με μεγάλη επιτυχία. Επίσης, προσπαθούμε να έχουμε μια μονοπευθυντική θηρίδα για τις μεταναστευτικές ροές και παρότι δεν λαμβάνουμε καμία χρηματοδότηση, έχουμε καταφέρει να καταγράψουμε 112.000 μετανάστες και πρόσφυγες το 2015. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε την κοινωνία των πολιτών, η οποία βοηθά πάρα πολύ στην διαδικασία ένταξης και προσπαθεί να επηρεάσει την ε, κοινή γνώμη και να αλλάξει τη στάση της απέναντι στη μετανάστευση. Επίσης, η ειρηνευτική διαμεσολάβηση. Όπως ξέρετε, η Βαρκελόνη έχει πληγεί από την κρίση, έχει υποστεί πολύ μεγάλες περικοπές του προϋπολογισμού της, ε, υποφέρει από ανεργία. Πήγαμε από το 7% στο 22% ανεργίας μέσα σε λίγα χρόνια. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και ποια πιστεύετε εσείς ε, πως είναι η άποψη των ε, πολιτών μας για τη μετανάστευση. Κάναμε μία έρευνα. Ρωτήσαμε τους κατοίκους τι αισθάνονται για τη μετανάστευση και τι πιστεύουν, ε, αν πιστεύουν ότι επηρέασε η, μετανά, η, κρίση, η μετανάστευση την κρίση και αντίστροφα. Σίγουρα οι κάτοικοι της Βαρκελόνης έχουν ε, προβλήματα, όμως η έρευνά μας συμπέρανε πως οι πολίτες μας δεν έριξαν το φταίξιμο ε, για την κρίση στους μετανάστες. Και πιστεύω λοιπόν πως τα αποτελέσματα της Βαρκελόνης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα εισήγηση. Προσπάθησα, αλλά δεν κατάφερα να σας ε, ε, διακόψω, αλλά ήθελα να σας ακούσω μέχρι το τέλος, οπότε για να δώσουμε τώρα το λόγο ε, στον κύριο Λανταβάσο, ο οποίος ε, έχει αναλάβει τα ζητήματα της ανάπτυξης στις πόλεις, της ανάπτυξης ε, στην Βόρεια Ευρώπη ως ε, ε, διευθυντής και είναι γενικός διευθυντής της Αρμόδιας Διεύθυνσης. Υπάρχουν θέματα που τα έχουν θέσει πολύ μέχρι τώρα. Ο κύριος Λανταμπάς, ο τρόπο να μας ενημερώσει όσον αφορά τις προτάσεις για το θεματολόγιο της πόλης από την Γενική Διεύθυνση της Περιφερειακής Πολιτικής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και σε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε ούτω ώστε να μπορέσω να μιλήσω σε αυτή την ενδιαφέρουσα ακρόαση. Ακούσαμε αυτά τα ζητήματα και μας δίνεται τον λόγο ε, τελευταίο στη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τα σκεφτούμε καλύτερα και για να ξεκινήσουμε από τα πιο στοιχειώδη ε, τι γίνεται και γιατί χρειάζεται. Χρειάζεται ένα πλαίσιο ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια αποτελεσματική πολιτική της ε, πόλης. Και για εμάς η πολιτική για τις πόλεις αφορά κάποιες πολιτικές οι οποίες θα είναι ολοκληρωμένες και θα έχουν τρεις άξονες ε, κοινωνική, κοινωνική ολοκλήρωση, καταπολέμηση της ε, ε και θα πρέπει να δούμε τώρα κατά πόσον έχουμε το νομικό πλαίσιο. Αυτά δεν ε, ε, αφορούν την συνθήκη. Όμως αυτό το οποίο έχουμε στη συνθήκη είναι η εδαφική συνοχή. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η ανάπτυξη να συνδέεται με την πολιτική των πόλεων και αυτό για μας ε, είναι μια βάση για να αναλάβουμε δράση. Και σας παραπέμπω στο ερώτημα γιατί χρειάζεται μια με ένα τέτοιο θεματολόγιο. Ε, θέλουμε να δούμε πώς είναι η κατάσταση στην πραγματικότητα στις πόλεις και θα πρέπει να από εδώ να κρυθεί επιτυχία ή αποτυχία. Γιατί εδώ ε, κρίνεται το πώς οι Ευρωπαίοι εκτιμούν αυτά τα οποία κάνουμε. Οπότε και θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή την ε, προσπάθεια για το θεματολόγιο. Είναι κοινή προσπάθεια με το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιών και τα κράτη-μέλη. Για να δούμε επομένω με συντομία ποια είναι η διάσταση που αφορά την πολιτική για τις πόλεις, ε, πολιτικές μας. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αν ρίξετε μία ματιά ε, στις λεπτομέρειες του προγράμματος εργασίας του 2015 θα διαπιστώσετε ότι εκεί γρητός αναφέρουμε όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρχει καλύτερη εταιρική σχέση με τις πόλεις και αυτές μας οι πολιτικές να είναι πιο αποτελεσματικές. Οι δε επιπτώσεις ε, να είναι πιο ουσιαστικές ε, και έτσι έχουν προσέξει και την τοπική διάσταση σε αυτό το πρόγραμμα εργασιών μας. Τώρα, γιατί πολιτική για τις πόλεις. Ε, Ανέφερε ο συμπρόεδρος και, και κάποιοι από τους ε, καθηγητές ότι έχουμε τα τρία τέταρτα του ΑΕΠ τα οποία εκεί γεννώνται και παράγονται αλλά έχουμε και επτά στις δέκα προτεραιότητες που έθεσε ο πρόεδρος Γιούνκερ επηρεάζουν ή μπορούν να πειράσουν σημαντικά το μέλλον και την ανάπτυξη των ε, πόλεων. Είναι κάτι σαν ευφυείς οι πόλεις ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη στις περιοχές όπου βρίσκονται αυτές οι πόλεις, αυτοί ας πούμε κόμβοι. Για να προχωρήσουμε λίγο ταχύτερα. Ποια είναι τα αποτελέσματα του, του θεματολογίου. Μπορούμε να δούμε διάφορα συστατικά που συναποτελούν αυτή την ε, πολιτική. Πάντως όσον αφορά το θεματολόγιο αυτό το οποίο έχουμε είναι εταιρικέ σχέσεις σε 12 θέματα. Και όλα αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη ε, λόγω της Ολλανδικής Προεδρίας. Οπότε βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι απτά και πρακτικά. Και πρόκειται για προγράμματα δράσης. Η διαδρομή θα είναι δύσκολη, αλλά θα είναι και διαδραστική. Αλλά όλα αυτά αποτελούν την ουσία του θεματολογίου μας. Όλα αυτά τα καθόρισαν οι εμπλεκόμενοι που κάθισαν και τα συζήτησαν. Είχαμε 12 στρογγυλές τράπεζες και αναπτύχθηκαν αυτά τα 12 προγράμματα δράσης. Οπότε όλα αυτά θα έρθουν το Μάη, κατόπιν θα κάτσουμε να δούμε τι έγινε. Ο κύριος Άλμπρεχτ επίσης ε, μας είπε ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την διαδρομή αυτή, να μάθουμε και τελικά όλα αυτά να τα ενσωματώσουμε στο μέλλον όταν έρθει η ώρα να κάνουμε την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Έτσι θα προχωρήσουμε, έτσι θα προσπαθήσουμε. Διακυβέρνηση τώρα, σε αυτή την διαφάνεια βλέπετε ότι η διακυβέρνηση ε, σημαίνει το ποιο κάθεται στο τραπέζι των συζητήσεων. Αλλά για εμά πάντω ε, είναι η ουσία μια από πολιτική η διακυβέρνηση. Και πολλοί έχουν μιλήσει για οριζόντια διακυβέρνηση και κάθε διακυβέρνηση. Οριζόντια σημαίνει ε, πολλούς εμπλεκόμενους, θα πρέπει να μην έχουμε ε, τεχνητούς ε, θεσμικούς φραγμούς και κάθετα αντίστοιχα σημαίνει ότι μια σωστή πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται σε μια καλή περιφερειακή πολιτική γιατί εδώ πέρα υπάρχει αλληλεπίδραση ξεκάθαρη άρα όλα αυτά είναι διακριτά αλλά διασυνδέονται. Τώρα για να δούμε ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο. Πέραν των όσων βλέπετε εδώ θεωρούμε ότι το πολιτικό πλαίσιο πρόκειται σύντομα να είναι ένα πλαίσιο αξιόλογο και πολιτικό στα πλαίσια του Συμφώνου του Άμστερνταμ. Και αυτό είναι η βάση της συνεργασίας μας, αλλά και με την Ολλανδική Προεδρία. Να υπάρχει επομένως σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, ώστε να προωθήσουμε την πολιτική για τις πόλεις. Και επομένως να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Οπότε για να γίνει κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε την στήριξη από εσά. Από ό,τι ξέρω ισχύει αυτό. Ξέρουμε τι έχετε κάνει, τι θα κάνετε, όπως και η Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Βεβαίω και για τους λόγους που προανέφερα ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ότι υπάρχει ένα project group από δύο αντιπροέδρους και υπάρχουν ε, συχνές συναντήσεις ε, διαφορετικών ε, επιτρόπων. Έχουμε τουλάχιστον 20 γενικούς διευθυντές οι οποίοι ασχολούνται με την υπόθεση αυτή και 6 με μια μονάδα που έχει σχέση με το θεματολόγιο με την Επιτροπή για τις Πόλεις. Οπότε όπως σας είπα, αυτό έχει να κάνει και με τις προτεραιότητες Juncker. Οπότε και θεωρούμε ότι έχουμε αυτά τα 12 θέματα προτεραιότητας. Αυτό είναι ανοιχτός κατάλογος ούτως υπήν. Οπότε αν κανείς θέλει μπορεί να προσθέσει ε, κάποια θέματα Αυτά δεν είναι τίποτα θέσφατα. Χρειάζεται να είναι κάτι το οποίο να βγάζει νόημα για τους ε, Ευρωπαίους. Και φυσικά χρειάζεται να υπάρχει συμφωνία επί τη διακυβέρνηση όπω είπαμε πριν. Τώρα για να δούμε τι γίνει μέχρι τώρα. Έχουμε τέσσερι εταιρικέ σχέσει. Είπαμε ότι η Ολλανδική κυβέρνηση έχει κάνει συνεδριάσει. Τελευταία συνάντηση αφορούσε του πρόσφυγε και ελπίζουμε ότι εδώ θα είναι πρώτο πόρο το Άμστερνταμ αλλά και ίσως άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ε, το Φεβρουάριο όλα αυτά θα προχωρήσουν. Επίσης ε, έχουμε και μια αξιολόγηση των επιπτώσεων, ε, κάποια σεμινάρια, επίσης και την ενεργειακή απόδοση σε κτίρια εκπομπέ διοξιδίου και αυτά και επίσης ε, αναπτύσσουμε αυτή την ε, πλατφόρμα δεδομένων για τι ε, πόλει για να ξέρουμε για το τι μιλάμε, κάποια κριτήρια, κάποιοι δείκτες και όλα αυτά γίνονται στο κεντρικό κέντρο ερευνών Επίση, καταγράφουμε τις προτεραιότητες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε συνέργειες, συμπληρωματικότητες, να κάνουμε ό,τι μπορούμε με τους δεδομένους πόρους. Και επίσης γι' αυτό έχουμε και την μοναπευθυντική θηρίδα One Stop Shop για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και περί τα τέλη του έτους ήδη κάτι να έχει προκύψει. Επίσης έχουμε τις ε, καινοτόμες δράσεις για τις πόλεις. Θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα δημιουργηθεί αυτό μέχρι τέλος Μαρτίου και έχουν διατεθεί 80 εκατομμύρια για τέσσερα ε, βασικά θέματα που συνδέονται με τα άλλα 12 του θεματολογίου, Αυτό το οποία σας ανέφερα, σας είπα για τους ειδούντες άσυλο και για τους πρόσφυγες. Αυτό είναι ένα από τα θέματα για κάποιες πόλεις των 50.000 επί τρία χρόνια, ε, θα πέσουν 5 εκατομμύρια, θα υπάρχει ένας ε, ανταγωνισμός ή ένας διαγωνισμός μάλλον θα υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτό είναι μόνο ο πρώτος διαγωνισμός έχουμε πάνω από 300 εκατομμύρια που έχουν διατεθεί και αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να δούμε ε, ποιος τι μπορεί να κάνει για να μπορέσουμε αυτά να πολλαπλασιαστούν και έτσι να ασχοληθούν για να μπλαγούν περισσότερες πόλεις τώρα. Τι γίνεται με το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, διότι πολλοί είπαν τι έχει γίνει. Ναι, νομίζω ότι από το 1994 έχουμε τόσες πόλεις που έχουν εμπλακεί τότε που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Σήμερα έχουμε 15 δις συνολικά στα χέρια των πόλεων. Έχουμε καινούργια εργαλεία. Μερικοί λένε ότι κάποια από αυτά είναι πολύ μπερδεμένα. Επομένως στον ψηφικό κανονισμό έχουμε τα καινούργια εργαλεία πολιτικής και για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει έναν περιορισμό ότι θα πρέπει οι ίδιες οι πόλεις να επενδύσουν μέχρι 15 δις στις πόλεις. Και για να δείτε όλο το ψηφιδωτό είπαμε ότι έχουμε πάνω από 100 δις τα οποία θα δαπανηθούν στις πόλεις και επίσης το κοινωνικό ταμείο πρόκειται για κοινωνική πολιτική να δαπανήσει. Έχουμε και το Urbact για την διάδοση της ε, γνώσης όσον αφορά την ε, άσκηση και χάραξη πολιτικής. Είπαμε ότι έχουμε τις καινοτομίες δράσεις, έχουμε το ίντερνετ και το ΕΣΠΟΝ. Οπότε βλέπετε κύριε Πρόεδρε ότι με λίγα λόγια, να πως έχει σήμερα η κατάσταση με το λόγια της πόλης. Βεβαίω κάνουμε πολύ περισσότερο πλευρά επιτροπής Επιτροπή, αλλά σα δίνουμε μια πρόγευση για το πώς θέλουμε εσείς να συμβάλλετε στην υπόθεση αυτή, Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο τελευταίος ομιλητής και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε με τη συζήτηση. Ο κύριο Κατάνεο. Σα ευχαριστώ κυρία Μιχαήλοβα. Τέσσερι μου έχουν ζητήσει το λόγο από την Επιτροπή των Περιφερειών. Πρώτο ηγητή, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μα δίνετε να δουλέψουμε πάνω στην ατζέντα για τα αστικά κέντρα και την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ απολύτω με τον κύριο Όλμπριχτ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητο να τονίσουμε τη σημασία που έχουν τα αστικά κέντρα και τη σημασία που έχει η συμμετοχή του στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής γιατί εκεί δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης και εκεί σφυριλατείται η συνοχή. Το έχω επαναλάβει. Και ε, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, δέσμευσης για να γίνει κάτι τέτοιο μετά από 20 χρόνια νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μια τομή. Η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολλά υποσχόμενη και ακριβής. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα όμως για να έχουμε δομική συμμετοχή των πόλεων στα τεκτενόμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αντίστροφα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε και να υποστηρίξουμε. Η Ευρώπη χρειάζεται την εξουσία των πόλεων για να φέρει αποτελέσματα και γι' αυτό δεν θα πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκή ατζέντα, αλλά για πολιτική για τα αστικά κέντρα αστική πολιτική. Και ο κύριος Όλμπριτ μας είπε ε, ότι θα πρέπει να γίνει μια αντιπαραβολή μεταξύ περιφερειακής πολιτικής και αστικής πολιτικής. Όμως στην Ευρώπη η πραγματικότητα έχει ως εξής. Όλο και περισσότερες πόλεις και περιφέρειες είναι ο χώρος όπου παράγεται κοινωνική συνοχή και δημιουργείται οικονομία. Η περιφερειακή πολιτική μπορεί να προσαρμόσει την αστική πολιτική και η αστική πολιτική μπορεί να διευρυνθεί στην περιφέρεια. Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί στην πράξη. Είναι κάτι που στηρίζω και ελπίζω να έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίπλα μας για να έχουμε ε, ε, εγγενώς δομικά ευρωπαϊκά εργαλεία, εγγενώς δομική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Και σε σχέση και με τους λοιπούς ομιλητές να πω ότι η ατζέντα για το άστι δεν αντιτίθεται στην Ήπεθρο. Αντίθετα ε, πρόκειται για συνδυασμό με την Ήπεθρο, για συνδυασμό με την περιφέρεια, για σύμπλευση. Ο σκοπός είναι να δούμε πώς χειριζόμαστε τις πόλεις μας η Ευρώπη, δεν πρέπει η Ευρώπη να διοικεί τις πόλεις. Εμείς το κάνουμε αυτό. Από μόνοι μας. Και σε σχέση με τον τρίτο μιλητή θα ήθελα να πω ότι ανέφερε αρχικά αστικά στοιχεία ε, ότι υπάρχουν όταν έχουμε ε, οικισμό κάτω από 300.000 κατοίκους. Το 65% του πληθυσμού στην Ευρώπη, ε, το 68% ζει ε, σε αστικά κέντρα και το μισό από αυτά ζει σε πόλεις που ο πληθυσμός τους δεν ξεπερνάει τους 100.000 κατοίκους. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς. Δεν, είναι, ε, δεν μιλούμε μόνο για τις μέγα πόλεις, τις μητροπόλεις, τις πολύ μεγάλες πόλεις. Μιλούμε για τις κανονικές πόλεις των 20.000, των 30.000 κατοίκων όπου πραγματικά είναι αστικά κέντρα. Είναι το κέντρο κάθε περιφέρειας. Εκεί ζουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και πρέπει να υπάρχει σωστή συνεργασία με ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν και δήμοι βεβαίω με 200.000 ανθρώπους, με 200.000 κατοίκους που στερούνται έργων υποδομής. Βλέπετε την ποικιλομορφία στην Ευρώπη ε, και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, να την αναδείξουμε αυτή την ποικιλομορφία και να πετύχουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ήπειρος να είναι επιτυχημένη και πρέπει να το κάνουμε τώρα, γιατί μέσα σε 25 χρόνια μόνο το 7% ε, του πληθυσμού παγκοσμίω θα ζει στην Ευρώπη και για να έχουν καλή θέση τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας πρέπει ήδη να ξεκινήσουμε τη δράση μας από τώρα. Ευχαριστώ κύριο Φανίτς Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τα δύο αυτά θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών. Και να υπενθυμίσω γιατί καθόμαστε δίπλα-δίπλα σε αυτό τον οδικό χάρτη πορείας προς το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Ακριβώς λόγω αυτού που είπατε εσείς πριν από λίγο. Ότι 20 χρόνια συζητούμε, έχει γίνει προεργασία. Όταν όμως ξεκίνησε η Ευρώπη με τον Τελόρ, ήταν η Ευρώπη των περιφερειών και όχι η Ευρώπη των πόλεων. Τι κάναμε λοιπόν. Ανοίξαμε την πόρτα, διευρύναμε την πολιτική αυτή έτσι ώστε να ανοίξει ένας διεύλος επικοινωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη μία και πόλεων από την άλλη. Αν δείτε τη νέα συνθήκη, κάτι έχει προσθεθεί και είναι η έννοια της εδαφικής συνοχής. Τελεία. Και αυτή είναι και η μόνη αλλαγή. Και εκεί ε, ε, υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω εξελίξεις μετά το 2020, αλλά υπάρχει και η παγίδα. Όσες πόλεις βρίσκονται σε ε, εκτάσεις εδερφικής συνοχής και μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική ευμερία, στην περαιτέρω συνοχή, θα δουν το ρόλο του αναβαθμισμένο. Πολλοί έχουν περάσει 30 χρόνια ασχολούμενοι με την περιφερειακή πολιτική. το ερώτημα που έχω να απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη και τα λεγόμενα του προηγούμενου ομιλητή, είναι το εξή. Ε, το πολυεπίπεδο διακυβέρνηση των πόλεων με την προστιθέμενη τους αξία, με τα προβλήματα και τις λύσεις που κομίζουν, ε, ε είναι το επίπεδο που μπορούμε να χαράξουμε πολιτική και να έχουμε εκεί μια ε, λεωφόρο επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα Ευρωπαϊκά Κονδυλία. τα τελευταία χρόνια, για να έχει κανείς περιφερειακά κονδύλια ως προϋπόθεση πρέπει να έχει ένα σχέδιο εξειδίκευσης των περιφερειών. Είναι το νέο στοιχείο. Απ' την άλλη με τη σύμβαση των δημάρχων είχαμε τις έξυπνες πόλεις. Ε, αϊφόρες, ε, ανέργεια κτλ. Αυτά τα δύο αναπτύχθηκαν με τελείως διαφορετικό τρόπο από τη μία γενική διεύθυνση στην άλλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να συνδεθούν οι πολιτικές και πρέπει να δούμε πώς ε, θα είναι το παραδοτέο μας, πού θα κάνουμε τα επόμενα βήματα. Και χαίρομαι διότι βλέπω ότι ακούει και το Συμβούλιο εδώ και είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε ποιο είναι το διαφορετικό. Το Συμβούλιο λοιπόν θέλω να μας πει σήμερα τι θέλει να κάνει. Θέλει να εμπλύνει μέσα εταίρους σε αυτό το σύμφωνο του Άμστερνταμ ή θα είναι μόνο μια συμφωνία αμυγό συμβουλίου εντό του Συμβουλίου των Κρατών Μελών, ε, δηλαδή με τον παραδοσιακό παλαιομοδητικό τρόπο. Το σύμφωνο του Άμστερνταμ θα είναι συμφωνία κρατών μελών υπουργών στο Συμβούλιο ή θα εμπλέξει και ε, δημάρχου και οργανωμένη κοινωνία των πολιτών ε, και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα νέο σημείο ισορροπίας. Τι θα είναι, θα είναι η δήλωση του Άμστερνταμ με άλλο όνομα, με άλλο κείμενο αν θέλετε ή γραμμένη σε διαφορετικό χαρτί ή θα είναι μαζί με π.χ. 150 συμφωνίες με εταίρους, ε, με πόλεις, με ε, οτάμε διαφόρους φορείς που θέλουν να ανέβουν σε αυτό το τρένο από τη στιγμή που μετά το 2020 θα έχουμε μεγάλες αλλαγές. Είναι μια πρωτοβουλία μιας νέας κοινή μοιρασμένη ευθύνη έχετε ένα μεγάλο φάκελο με συμφωνίες ε, που έχετε ήδη πετύχει εσείς με διάφορες πόλεις και μέλη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών για το σύμφωνο του Άμσεντα Ή θα είναι μια συμφωνία παραδοσιακή τύπου Συμβουλίου. Θα σταματήσω κάπου εδώ γιατί θέλω να μάθω πόσο ικανοποιημένοι θα είμαστε το Μάιο με την υπογραφή του συμφώνου αυτού η Πρόεδρος. Ενδιαφέρουσες προσδοκίες έχετε για το τι μπορεί να σας κάνει ευτυχισμένο το Μάιο. Ας θα ακούσουμε ε, από τον Συμπρόεδρο. Θα ακούσουμε από την Ολλανδική Προεδρία αργότερα. Ο κύριος Κατάνεο, επόμενος ομιλητής από την ε, Επιτροπή των Περιφερειών. Η κυρία Τάνκερ Λόπες. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνω την ε, δυσαρέσκεια που επικρατεί στην αίθουσα, διότι πρόκειται για μια αποτυχία της πολιτικής τα τελευταία 20 χρόνια πρέπει να δούμε τι έπρεπε να κάνουμε, τι στόχους είχαμε και να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι δεν έγιναν πολλά. Όμως πιστεύω πως ε, δεν ε, πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά το αντίθετο. Έχουμε καταφέρει να έρθουμε σε μια αμοιβαία συνεννόηση, να καταλήξουμε στις ε, σημαντικές για εμάς προκλήσεις. Πρέπει να πορευτούμε προς την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών στόχων και να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από τις υφιστάμενες δυνατότητες και οι πόλεις επίσης δεν πρέπει να διαχωρίζονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες ως προς την συμμετοχή τους και τη συνεισφορά τους στο αστικό θεματολόγιο. Το σύμφωνο του Άμστερνταμ ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προς ε, μια αστική πολιτική την οποία πρέπει να συνοδεύσουμε και εμείς. Μία πολιτική η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική, καλύτερη νομοθεσία, δηλαδή καλύτερη χρηματοδότηση, καλύτερο συντονισμός. Δεν είναι μία νέα νομοθετική πρόταση, αλλά η υλοποίηση ε, και η καλύτερη χρήση των μέσων που ήδη υπάρχουν. Αυτό που φάνηκε από αυτήν την ε, παρουσίαση, από όλε τις παρουσιάσεις, είναι ότι πραγματικά χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό. Κάτι το οποίο αναγράφεται και στο σύμφωνο του Άμστερνταμ. Πιστεύω όμως πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι πιστεύω πως δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο εάν οι γενικές διευθύνσεις μεταξύ τους δεν συνεργάζονται με τρόπο επικοδομητικό. Και εδώ πιστεύω πως πρέπει πράγματι να ε, έχουμε έναν ε, συντονιστή, έναν συντονιστή πολιτικό, ο οποίος θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, καλή συνεργασία. Αυτό θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία και το πρόγραμμα εργασίας μας τα επόμενα χρόνια. Υπόθηκε στην αρχή, στα πλαίσια της ε, σε εδαφικής συνοχής και των ε, θεμελίων αυτής, ότι το σύμφωνο του Άμστερνταμ πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα βασικό θεμελιώδες κείμενο, ε, ως, που θα βοηθήσει στην έβρεση μιας μεθόδου εργασίας και πιστεύω πως ορισμένα στοιχεία, ορισμένα στοιχεία από το σύμφωνο του Άμστερνταμ πρέπει να τονιστούν. Πρέπει να τονιστεί για παράδειγμα ο δεσμευτικός χαρακτήρας έτσι ώστε να μην καταλήξουμε ε, μερικά χρόνια αργότερα να πούμε ότι πολύ ωραία τα είπαμε αλλά δεν έγινε τίποτα. Όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά πρέπει ε, να τονιστεί οπωσδήποτε ότι χρειάζεται διαφάνεια. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και επίσης χρειάζεται η συμμετοχή όλων των φορέων. Και τώρα θα περάσω και σε ένα άλλο σχόλιο, σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και νομίζω δεν αναφέρθηκε αρκετά. Σίγουρα ε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. ταρτίζουμε τριετή σχέδια, μετά περνάμε από μία περίοδο αξιολόγησης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι χρειάζεται διαφάνεια και στην υποβολή εκθέσεων και στο σύστημα αξιολόγησης. Γι' αυτό χρειάζεται μια τακτική παρακολούθηση, τακτικός έλεγχος, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε αυτά που ε, ζητούνται, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη νέα διαρθρωτική περίοδο και να ε, δημιουργήσουμε μια λευκή βίβλο η οποία θα ε, αποτελέσει βάση για τις περαιτέρω εργασίες μας. Όχι κάθε τρία χρόνια, αλλά κάθε ενάμιση χρόνο αξιολόγηση. Αυτή είναι η άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών μέσα από τη γνωμοδότησή της και ελπίζω να βρει μεγάλη απήχηση σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Το λόγο στα μέλη σας. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ριπαρό. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αυτά που ήθελα να πω ήδη τα ανέφεραν προηγούμενοι ομιλητές. Είναι πολύ σημαντικό για μια συνολική και ολιστική προσέγγιση να ακούμε για τις διπουργικές συναντήσεις και για τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν τις αστικές πολιτικές. Άλλωστε το άστι συνδέεται πάντοτε με την ενδοχώρα θα είναι επιτυχημένη αστική πολιτική εάν ε, συνάδει με την ενδοχώρα. Πολλοί ακούσαμε την ε, ιστορία επιτυχίας του Μπιλμπάου, πώς έβγαλαν 100 εκατομμύρια ευρώ με το Μουσείο Guggenheim. Αλλά δεν γίνεται λόγος για τα 100 εκατομμύρια ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για τα συστήματα οδικών μεταφορών και άλλων μεταφορών που συνέβησαν το, το Μπιλμπάου με τις άλλες περιοχές και πόλεις. Αυτό είναι μια ιστορία επιτυχίας δεν είναι η ίδια περιφέρεια. Επεκτείνεται με την επέκταση του συστήματος μεταφορών. Επεκτείνεται η περιφέρεια με τη συνεργασία των μεταξύ των διαφόρων και διαφορετικών πόλεων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και σημαντικό είναι να δούμε πώς συνεργάζονται οι πόλεις για να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Δημιουργείται μια διαδικασία εκεί και στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται και τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, τα οποία δεν έρχονται στη συνέχεια εκ των υστέρων να αξιολογήσουν και να μελετήσουν το τι συνέβη, αλλά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κομίζουν την ε, πολυπραγμοσύνη τους. Και εάν τα καταφέρουμε, αν καταφέρουμε αυτό να κάνουμε και να εμπλέξουμε όλα τα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης από το ευρωπαϊκό μέχρι και το τοπικό, τότε σίγουρα θα μας ικανοποιήσει το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Μιχάλοβα. Ο κύριος Κατάνα. Η κυρία Φανέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε συμπρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή την τόσο χρήσιμη συζήτηση. Ε, πολύ συγκεκριμένη. Ας ευχηθούμε γιατί ξεκινώ από τη δική μου χώρα. Γιατί χρειάζεται ένας προγραμματισμός των 28 χωρών μελών και έτσι να κατευθυνθούμε προς το αστικό πρόγραμμα. Μιλούμε για ένα δις το ίμιση από τα διευθυντικά ταμεία. Και έτσι να έχουμε αυτόν τον κύκλο προβληματισμού και έτσι να προσπαθήσουμε να έχουμε μία παρέμβαση στις 13 μεγαλύτερες μας πόλεις και ξεκινώ με την πεποίθηση ότι αυτό το θεματολόγιο έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο για τα κράτη-μέλη και επομένως να είναι ξεκάθαρο που, ε, ποιος έχει την αρμοδιότητα και τι, έχει, τι, έχουν τα κράτη-μέλη, τι έχουν οι πόλεις, τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε σε επίπεδο κρατών μελών να προχωρήσουμε και να καινοτομήσουμε ακόμα και στο επίπεδο του προγραμματισμού με κάποια λειτουργικά, ψηφιακά προγράμματα εθνικά που να αφορούν τις αστικές περιοχές. Πρόκειται για ένα σημείο όπου νομίζω ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε, να, να, στα πλαίσια αυτής της ε, προβληματικής που τώρα συζητούμε οπότε και έτσι να έχουμε περισσότερες δυνατότητες και έτσι να μπορούμε να ε, διασυνδέσουμε αυτά τα θέματα και να διαμορφώσουμε μια πραγματική πολιτική πλευρά του θυμητολογίου και έτσι θα πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, παράλληλα με τις περιφερειακές πολιτικές κάποιες πολιτικές ε, τοπικές. Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μια αλλαγή εκβάθρων και έτσι να έχουμε τελικά κάποια κριτήρια ε, οικονομικά να, υπάρχει, να υπάρχουν οικονομικοί πόροι και να δούμε τι γίνεται στο ιστορικό των χώρων μελών και να μπορέσουμε επίσης να αποτιμήσουμε τι γίνεται σε επίπεδο διακυβέρνησης και σε επίπεδο επιδόσεων. Επίσης, ε, μπράβο για την επιλογή των θεμάτων που έχουν επιλεγεί, διότι έχουμε προτεραιότητα την μετανάστευση αλλά και την φτώχεια, οπότε και εγώ είμαι πεπισμένη ότι όλα αυτά τα οποία εδώ καλύπτονται είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εμπνεύσουν τις διάφορες πλευρές της πολιτικής μας, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ανάπτυξη και σε βιώσιμη ανάπτυξη ε, και όσον αφορά τα ψηφιακά. Οπότε ε, θα πρέπει αυτό να είναι οι βασικές μας επιλογές και προτεραιότητες. Να πάει προς τα εκεί η Ευρώπη για τα ε, θέματα που θέλει να φροντίσει. Τώρα τελευταίο και σημαντικό θα πρέπει να τολμήσουμε ε, ούτως ώστε στην ε, καρδιά αυτού του, του ε, οράματος να έχουμε 4-5 προσπάθειες και καινοτόμες και θα πρέπει να δούμε τι είναι η συμμετοχική οικονομία, τι μπορεί να κάνουν οι πόλεις, τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών και πώς συμβαίνουν κάποια, κάποια, κάποια στοιχεία, πώς αναπτύσσονται κάποια που συμβαίνουν σε κάποια μέρη και όχι αλλού. Επομένως θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιες απόπειρες, να υπάρχει καινοτομία, να έχουμε αφετηρία τις άρεστες πολιτικές και να έχουμε επομένως έτσι μία προστιθέμενη αξία με αυτό το θεματολόγιο και να προκύψει συγκεκριμένη πολιτική ούτως ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να αλλάξουμε το πρόσωπο της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να αξιοποιήσω την ευκαιρία ε, της παρουσίας του εκπροσώπου του Συμβουλίου για να σας πω ότι έχετε θέσει ένα ερώτημα προς την Ολλανδική Προεδρία. Κύριε Κόλπα, έχετε το λόγο. Για μια πολύ σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Το πιο δύσκολο είναι αυτό, να είμαι σύντομος. Okay. Perhaps I, should sit now. Πάει και το πρώτο μου λεπτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης και ε, την Επιτροπή Ρέτζη ευχαριστώ και την Επιτροπή Κοτέρ. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η ακρόαση και εξαιρετικά σημαντική και έρχεται ε, σε, στην πιο κατάλληλη χρονική στιγμή θα έλεγα. Σημείωσα, εάν δεν απατώμε, ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα εντός της εθούσης. Όχι μόνο ε, από τα μέλη της Επιτροπής Κοτέρ και της Επιτροπής Ρέτζι, αλλά και οι ομιλητές εξέφρασαν την ελπίδα τους και αυτό είναι σημαντικό. Όλοι είπαν ότι το σύμφωνο του Άμστερνταμ ε, φέρνει ελπίδα. Είπατε όμως ότι έχει σχέση με τις λέξεις και πράγματι ε, κάθε σύμφωνο αποτελείται από λέξεις. Είναι όμως κάτι παραπάνω από αυτό. Ε, είναι ένα κάλεσμα στις πόλεις και στα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στην ατζέντα Juncker. Πιστεύουμε ότι για να πετύχει η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί ενεργά με τις πόλεις και τις περιφέρειες. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Βέστφαλ, την εισηγήτρια, για αυτή την έκθεση για την αστική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται μόνο λόγος για την, εδαφ... για την πολιτική συνοχής. Γίνεται λόγος και για την πολιτική την αστική. Για το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην ατζέντα Juncker και στις 7 από τις 10 προτεραιότητές της. Αυτό το οποίο σημειώνω είναι ότι ήδη υπάρχει δυναμισμός. Ε, ξεκινούν αστικές εταιρικές σχέσεις. Ε, γίνεται συζήτηση για αστικές καινοτόμε δράσεις, τις οποίες διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αρμόδια γενική της διεύθυνση. Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ ενεργή και δραστήρια εντός της Κομισιόν. Ε, πηγαίνει στους συνομιλητές και λέει ξεχάστε ε, τα μεμονωμένα. Χρειαζόμαστε ενιαίες και ολοκληρωμένες πολιτικές. Έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην ατζέντα Juncker. Επομένως, βλέπετε ότι υπάρχει μια κάποια καινοτομία και αυτό το οποίο θέλει η Ολλανδική Προεδρία να πετύχει το Μάιο είναι η παγίωση όλων αυτών. Ε, η παγίωσή τους με επιστέγασμα την επικύρωσή τους σε υπουργική διάσκεψη στο Άμστερνταμ και τα κράτη-μέλη επιθυμούν να εμπλακούν, να συμμετάσχουν σε αυτή την πολυεπίπεδη διαδικασία. Δεν είναι μια διαδικασία την οποία οδηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο ή το Συμβούλιο μόνο. Είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία και χρειαζόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη και των πόλεων και των περιφερειών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι θετικά τα κράτη-μέλη σε αυτή την εξέλιξη. Εγώ το ελπίζω και το πιστεύω και αν όντως ισχύσει αυτό και είναι θετικά τα κράτη-μέλη θέλουμε αυτό να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στα τέλη Ιουνίου με την, με την έννοια της δήλωση βεβαίως αλλά δήλωση από το Συμβούλιο. Αυτή είναι μια νέα προσέγγιση και γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Ο κ. είδε είπε ότι Όλοι και 20 γενικοί διευθυντέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δουλεύουν με τι πόλεις και για τι πόλει. Πολλέ φορέ δεν το ξέρουν, δεν το λαμβάνουν υπόψη του. Και κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει σε όλους τους τομείς και σε όλες τις διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως σε πολλές από τις γενικές διευθύνσεις υπάρχουν τμήματα για τα αστικά ε, κέντρα. Και η ομάδα του κ. Λαντεμπράσελ εργάζεται για να συνεργαστούν όλοι αυτοί. Και να απευθυνθούν και στον κύριο Τίμερμανς για καλύτερη νομοθεσία. Γιατί τελικά αυτό χρειαζόμαστε, καλύτερη νομοθεσία για να πετύχουμε αυτά τα οποία επιθυμούμε. Αυτά ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Η Συμπρόεδρος, ήσασταν αρκετά σύντομος και εγώ σας ευχαριστώ. Και μας παρουσιάσατε και πολλές πληροφορίες και πολλά στοιχεία. Ο κύριος Κατάνεο. Θα ήθελα τώρα να στραφώ προς τους ομιλητές και να τους ρωτήσω. Έχετε παρατηρήσεις καταληκτικές πριν τα συμπεράσματα those speakers who some... Θα ήθελε κάποιος να κάνει κάποια παρατηρήση, κάποιο σχόλιο. Παρακαλώ. Ναι, δεν ήθελα να είμαι αρνητικό, απλά να προκαλέσω. Και πιστεύω πω προκαλέσα το σωστό αποτέλεσμα. Πιστεύω πω ε, το κείμενο αυτό που βλέπω είναι ό,τι καλύτερο έχω δει τα τελευταία χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρήσουμε τι υποσχέσει μα. Αυτό λοιπόν είχα να πω και δεν είμαι απεσιόδοξο. Το αντίθετο, ε, έχω πολλέ ελπίδε. Σα ευχαριστήσω πολύ. Κυρία Άμσα, ευχαριστώ. Να σας πω πως πρόσφατα τελείωσε μία εκ των υστέρων αξιολόγηση διάφορων αστικών έργων που περιλαμβάνονται στα αστικά ε, στα διαστατικά ταμεία. Εσείς είπατε πως πρέπει να μάθουμε από τις αξιολογήσεις, όμως ε, δεν τις διαβάζουν και πολύ. Και αυτό θα έπρεπε να μας λέει κάτι για το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επηρεάσει αυτές τις δράσεις από τη βάση προς τα πάνω ή και να μην τις επηρεάσει. Ναι, θα είμαι σύντομος. Θα έλεγα ότι το αστικό θεματολόγιο φυσικά και είναι ευπρόστεκτο και αυτό το λέω σε κάποιος που εργάζεται για τις πόλεις, με τις πόλεις. Όμως είναι πολύ σημαντικό να είμαστε και ρεαλιστές. Η Ευρώπη αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούν και οι πολιτικές σε αυτήν την αλλαγή. Ιδιαίτερα οι πολίτες και τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει και πρέπει να γίνουν ε, πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη και των δύο επιτροπών και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κατάνεο για τα καταληκτικά σχόλια της συνεδρίασής μας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μιχαήλοβα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους για τις παρουσιάσεις τους, τις προκλητικές παρουσιάσεις, τα μέλη της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Κοτέρη της Επιτροπής των Περιφερειών για την ενεργό συμμετοχή τους. Θα ήθελα να τονίσω τα εξής τρία. Καταρχάς το Ευρωπαϊκό Αστικό Θεματολόγιο, κατά την άποψή μου, πρέπει να αφορά όλες τις αστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Φερκέρκ σε αυτό. Η Ευρώπη διαφέρει από τις υπόλοιπες υπήρους και η παρέμβαση του κύριου Έρμαν μας δείχνει ακριβώς αυτό. Η Ευρώπη είναι γεμάτη από μικρές αστικές περιοχές και δεν υπάρχουν τεράστιες μεγάλου πόλεις ή έστω πολύ λίγες. Υπάρχουν αντίθετα πολλές μεσαίου μεγέθους και μικρές πόλεις. Το αστικό θεματολόγιο λοιπόν πρέπει να αδεκτατροπτρίζει την δική μας αστική διάσταση και τις δικές μας συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη. Επίσης, χρειαζόμαστε ένα αστικό θεματολόγιο από τη βάση προς τα επάνω. το οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις πόλεις, τις περιφέρειες, τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση των πολιτικών. Και η εμπειρία μας δείχνει ότι η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες τοπικές αρχές, στα διάφορα επίπεδα διοίκησης, είναι κάτι που ε, βοηθά πάρα πολύ. Η συνεργασία λοιπόν είναι σημαντική και όχι ο ανταγωνισμός. Και τέλος να πω πως συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Όλμπριχτ. Χρειαζόμαστε όχι αστικό θεματολόγιο, αλλά αστικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύμφωνο του Άμστερνταμ και το αστικό θεματολόγιο που ήταν και το επίκεντρο της συζήτησής μας σήμερα πρέπει να στοχεύει στην καλύτερη βελτιωμένη ευρωπαϊκή αστική πολιτική. Ελπίζω λοιπόν να είμαστε στη θέση να συμμετάσχουμε έτσι ώστε να βελτιωθεί το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Διάβασα το προσχέδιο, το οποίο είναι ήδη μια πολύ καλή αφετηρία, όμως πιστεύω ότι το δεύτερο και τρίτο προσχέδιο θα πρέπει να είναι ακόμα πιο βελτιωμένα με καλύτερη αστική πολιτική και συγκεκριμένα μέσα για τους πολιτικούς, για τους πολίτες, για τους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή αστική πολιτική, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ζωής στις πόλεις και για τους πολίτες. Και αυτός πρέπει να είναι και ο τελικός μας στόχος και πιστεύω πως ε, αυτή είναι η καλή μέθοδος ε, η οποία θα μας οδηγήσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, πολύ κυρία Μιχαήλωβα και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να ανταλλάξουμε απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω κάποια Τελευταία λόγια, αγαπημένα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη, αγαπημένα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, κυρία Κατάνα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους και τους ομιλητές σήμερα για τη συμμετοχή τους στην συζήτηση. Έχουμε όλη επίγνωση ότι η Ευρώπη μεταβάλλεται εδαφικά και αντιμετωπίζει ένα άνευ προηγουμένου ε, νέο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Οι πόλεις και οι αστικές περιοχές είναι εκολαπτήρια καινοτομία και θα μας δώσουν μία χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη. Ας μην ξεχνάμε πως εμείς χαράσουμε πολιτική και Επομένως έχουμε μεγάλη ευθύνη για την εφαρμογή του αστικού θεματολογίου. Πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και να δημιουργήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των πολιτών στην Ευρώπη. Για πάνω από δύο δεκαετίες συζητούμε για την νέα αστική διάσταση και για τις πολιτικές που θα μας οδηγήσουν σε αυτήν. Είχαμε έναν αριθμό δηλώσεων και κειμένων. Ωστόσο, Πρέπει να σταματήσουν οι συζητήσεις. Έχει έρθει η ώρα η εταιρική μας σχέση να υλοποιηθεί και τα έργα μας να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις. Πιστεύω στην φιλόδοξη προσέγγιση, σε μια προσέγγιση που θα μας φέρει πιο κοντά στους στόχους της Ευρώπης 2020 για τους ανθρώπους στις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και πιστεύω πως η σημερινή συνεδρίαση ήταν μια καλή αρχή. Θα ήθελα να τονίσω μερικά στοιχεία. Καταρχάς, πιστεύουμε πως η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής πρέπει να ενισχυθεί. Η επερχόμενη αναθεώρηση της θετικής 2020 μας προσφέρει μια ιδανική ευκαιρία να επανέλθει η έμφαση στην αστική πολιτική. Έπειτα πιστεύουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέες μεθόδους για να βελτιώσει τη συνοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών και τις συνέργειες ανάμεσα στις εθνικές και περιφερειακές προσπάθειες. Είναι σαφές σήμερα ότι ο αυξανόμενος αριθμός των ε, πρωτοβουλειών που έχουν ως ε, στόχο την αστική πολιτική ε, αλληλοπικαλύπτονται και εμποδίζουν την δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται συνεκτίμηση των επιμέρους πολιτικών στην γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική, κάτι το οποίο συζητήσαμε και σήμερα. Και σε αυτά τα πλαίσια καλωσορίζουμε την συμπερίληψη των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση και στην χρήση των πολιτικών, κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο στις πόλεις μας. Όπως υπόθηκε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες κατάρτισης πολιτικής που θα έχει από τα αποτελέσματα. Επίσης, η απλούστευση πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του αστικού θεματολογίου. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές μας θα μειώσουν το διοικητικό άχθος και θα βοηθήσουν τις τοπικές και περιφερειακές ορχές να ε, τηρήσουν τις ε, υποσχέσεις τους. Πρέπει επίσης να συνδυάσουμε πόρους με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο και να διασφαλίσουμε, τους... διασφαλίσουμε έργα τα οποία θα οδηγήσουν σε πραγματικό όφελο στην κοινωνία και τους πολίτες. Και κλείνοντας, Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή η χρονιά θα είναι η αρχή μιας αποτελεσματικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Αστικού Θεματολογίου και της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Αστικής Πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτήν την ακρόαση και θα ήθελα εδώ να κλείσω την συνεδρίαση και να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής ότι η επόμενη τακτική συνεδρίαση θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου το απόγευμα και στις 16 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς εκ μέρους όλων σας. Σας ευχαριστώ. Λίγη συνεδρίαση.